Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος της Επιτροπής μας αφορά την πρόσφατη δήλωση της Ευρωπόλη σχετικά με τα 10.000 αγνοούμενα παιδιά μεταναστών. Όπως γνωρίζετε, ε, αναφέρθηκε σε πολλές εφημερίδες και γι' αυτό επιλέξαμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό σήμερα. Έχουμε καλέσει ε, εκπρόσωπους από την Ευρωπόλη κύριος ε, Νόιμαν την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, έχουμε την κυρία Δημητροπούλου και εκπρόσωπο από τη μη κυβερνητική οργάνωση Missing Children Europe, τον, την κυρία Μοράλης. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που ήρθατε σήμερα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους προσκεκλημένους μας και θα σας παρακαλέσω να μιλήσετε 8-10 λεπτά έκαστος. Έπειτα θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής και ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Νόημαν, εκπρόσωπο της Ευρωπόλ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, τους τελευταίους μήνες υπήρξαν δύο περιπτώσεις όπου θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε κάνει λάθος τις εκτιμήσεις μας. Την πρώτη φορά ο διευθυντής μας, ο κύριος Wainwright, μας είπε φέτος τον Ιανουάριο ότι η επόμενη τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη θα είναι άμεση. Και μόλις δύο μήνες αργότερα είχαμε τις επιθέσεις εδώ στις Βρυξέλλες. Η δεύτερη φορά ήταν όταν τον Ιανουάριο φέτος η Ευρωπόλ δήλωσε ότι υπάρχει πρόβλημα με αγνοούμενα παιδιά και τρεις μήνες αργότερα η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι πράγματι περίπου 5.000 ανήλικοι μετανάστες και πάνω από 400 ε, έφηβοι πάνω από 15 χρονών αγνοούνταν. Το φαινόμενο των αγνοούμενων παιδιών είναι πολυδιάστατο και παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Καταρχάς έχουμε φυσικά την, ε, το θέμα της ε, καταγραφής. Πιστεύω ότι ο αριθμός των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνευ προηγουμένου και πολλές φορές ε, οι εθνικές αρχές είναι υπερφορτωμένες, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην πρόκληση. Τώρα φτάνουν οι πρώτες ενδείξεις για το εύρος του προβλήματος και για ε, πρώτη φορά μας επιβεβαίωσε ένα κράτος μέλος, το πρώτο κράτος μέλος, ότι περίπου 5.000 ανήλικοι καταγράφηκαν ανάμεσα στο 2015 μέχρι σήμερα, αγνοούνται. Τους επόμενους μήνες και τις επόμενες ε, εβδομάδες αναμένουμε και άλλες εκθέσεις από άλλα κρατημέλη σχετικά με αγνοούμενους ασυνόδευτους ανήλικους. Έπειτα υπάρχει και το θέμα του τι κάνουμε με τις πληροφορίες που έχουμε. Καταρχάς, σύμφωνα με την είπατε αρμοστία του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες, περίπου 20% των μεταναστών που φτάνουν στην Ευρώπη από το 2015 μέχρι τώρα ήταν ανήλικοι, δηλαδή το 1 τρίτο περίπου. Κάτι το οποίο αποτελεί πολύ μεγάλο αριθμό φυσικά. Έπειτα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι μετανάστες βρίσκονται εκτεθειμένοι στις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Εκτιμάται ότι πάνω από 90% των μεταναστών χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτές οι ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος για να φτάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, ε, υπεύθυνοι για αυτές τις ομάδες είναι δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πολλές από αυτές τις ε, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που προσφέρουν αυτές τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δραστηριοποιούνται επίσης και ε, στον χώρο της διακίνησης ανθρώπων. Φυσικά υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί από αυτούς τους ανήλικους θα πέσουν θύματα διακίνησης ανθρώπων. Οι περισσότερες περιπτώσεις διακίνησης ανθρώπων που ε, φτάνουν στα χέρια μας έχουν να κάνουν με σεξουαλική ε, εκμετάλλευση και το φαινόμενο αυτό έχει ε, αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα ανήλικα θύματα του τράφικινγκ τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα, εμπλέκονται σε σεξουαλική εκμετάλλευση, απάτη σχετικά με τα επιδόματα και επαιτία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων, από όσο γνωρίζουμε, είναι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Τα παιδιά, οι ανήλικοι, θεωρούνται εμπόρευμα, εμπορεύσιμο είδος από αυτές τις ομάδες. Είναι εύκολο να μετακινηθούν ως υπήκοοι της Ένωσης από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, Υπάρχουν ανησυχίες ότι ανήλικοι μετανάστες ενδέχεται να γίνουν στόχος εκμετάλλευσης. Ακριβώς επειδή ε, είναι ανήλικοι, ευάλωτοι και χωρίς οικονομικούς πόρους. Αυτό που μπορώ λοιπόν να πω στην Επιτροπή σας σήμερα είναι ότι δυστυχώς πρέπει να επαναλάβουμε τις ανησυχίες μας για την παρούσα κατάσταση και επιβεβαιώνουμε την ε, μεγάλη πιθανότητα να γίνουν αυτοί οι ανήλικοι θύματα ε, αυτών των εγκλημάτων. Τώρα, από την πλευρά της επιβολής του νόμου, το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε είναι ότι η πλειοψηφία αυτών των ανήλικων θα ε, γίνουν λία αυτών των ε, ομάδων. Θα γίνουν λία του οργανωμένου εγκλήματος και αντικείμενα εκμετάλλευσης. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί από πολλές πτυχές. Καταρχάς, ε, οι αρχές επιβολής του νόμου πρέπει να ε, συζητήσουν τη συνδρομή της Ευρωπόλ για να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή και Ίσως θα έχετε συζητήσει τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης. Δεν θα επαναληφθώ λοιπόν, αλλά φυσικά θα χρειαστεί να ε, καταγραφούν οι ανήλικοι στα κράτη-μέλη στα οποία φτάνουν, κάτι το οποίο θα, μας, θα μπορέσει να μας δώσει μια εικόνα ε, του αριθμού τους και για να εκτιμήσουμε την έκταση του προβλήματος. Έπειτα χρειάζονται τα κατάλληλα συστήματα όπως ε, το σύστημα πληροφοριών Schengen, SIS, το οποίο θα επιτρέψει την καταγραφή των μεταναστών μέχρι 14 ετών το Eurodac, το οποίο θα επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων για να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν κάποιος ανήλικος που είναι καταγεγραμμένο σε ένα σύστημα υπάρχει και σε άλλο και εάν μπορούμε να βρούμε το που ε, βρίσκεται γεωγραφικά. Έπειτα, κάτι άλλο που έχει συζητηθεί στα νομοθετικά ε, σώματα και θα σας λέω κάτι καινούριο, αλλά για μας είναι η πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε τους ε, διαθέσιμους πόρους του συστήματος πληροφοριών Schengen έτσι ώστε να μπορούμε συστηματικά να διασταυρώνουμε τις ε, πληροφορίες που έχουμε για τους αγνοούμενους, για ε, τους ανήλικους, που με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε αποτελέσματα. Τώρα, πώς θα ευαισθητοποιήσουμε το κοινό έχουμε σκεφτεί πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να τραβήξουμε την προσοχή του κοινού. Οι εμπειρίες μας με, του, με τη, τον κατάλογο των καταζητούμενων στη συνιστοσελίδα μας είχε θετικά αποτελέσματα. Τους τελευταίους μήνες που είναι στο διαδίκτυο συναντήσαμε περίπου 10 περιπτώσεις ε, κατά τις οποίες μπορούσαμε να εντοπίσουμε και πιθανώς να μπορούμε να συλλάβουμε υπόπτους. Αυτό ίσως θα συνεισφέρει στην διαφάνεια της ε, κατάστασης. Επίσης, ε, πρέπει να συζητηθεί και το θέμα της γρήγορης ανταπόκρισης των αρχών επιβολής του νόμου. Υπάρχει ένας καλός μηχανισμός εμά που μας επιτρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Ήδη το πράττει αυτό η Ευρωπόλ ε, στην... στο χώρο της ε, διακίνησης ανθρώπων και τα δεδομένα που λαμβάνουμε τα επεξεργαζόμαστε και τα αποστέλουμε ξανά στα κράτη-μέλη. Επίση, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει και διεθνεί οργανισμοί συνεργάζονται μαζί μα για να, για να χρησιμοποιήσουμε βέλτιστε πρακτικέ. Τώρα, το πρόβλημα των ανήλικων προσφύγων είναι επίσης υπαρκτό και αρκετά μεγάλο. Ε, τι μαθαίνουμε από τις αρχές επιβολής του νόμου, πως είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα. Δεδομένου ότι οι ανήλικοι πρόσφυγες διακινούνται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων, είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Η Ευρωπόλη επιθυμεί να στηρίξει τις έρευνες και γι' αυτό ζητάει τη δική σας συνδρομή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Νόημαν. Ευχαριστώ. Τώρα, το λόγο στην υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Όσον αφορά τις διευκολύνσει υποδοχή ε, παιδιών, έχει πρόβλημα και αυτό το ξέρουμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ήδη από το 2009. Έχουμε υπογραμμίσει τον κίνδυνο κατάχρησης και κακοποίησης των παιδιών. Έχουμε αναφέρει το θέμα των αγνοούμενων ε, παιδιών σε νέα χώρες μέλη και όσον αφορά τα βιομετρικά δεδομένα, εμείς κοιτάμε κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μέσο για να εντοπιστούν αγνοούμενα ασυνόδευτα παιδιά. Θέλουμε οι αρχές προστασίας των παιδιών να μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες. Πόσα παιδιά είναι αγνοούμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και από πού. Δεν γνωρίζουμε τα ακριβή νούμερα. Τα έχουμε ακούσει από τον κύριο Νόημεν, από την ε, Europol αυτά. Και ακριβώς επειδή δεν το γνωρίζουμε, πρέπει να είναι κατανοητό ποιο και πού πρέπει να λέει και να ενημερώνει για κάθε φορά που αγνοείται ένα παιδί. Οι εθνικές αρχές πρέπει να ενημερώνονται που θα πρέπει να ενημερώνουν την αστυνομία. Και οι γονείς βέβαια πρέπει να κάνουν το ίδιο εννοείται. Συγγνώμη δεν γίνεται αυτό. Οπότε, υπάρχει ένας άγνωστος αριθμός αγνούμενων παιδιών που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ και μπορεί να είναι αγνούμενα αλλά δεν το ξέρουμε γιατί αφού δεν έχει καταγραφεί πουθενά. Δεύτερον, υπάρχουν παιδιά που έχουν καταγραφεί δύο φορές, σε δύο σημεία. Οπότε κάποια από τα, τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε συμπεριλαμβάνουν παιδιά ε, τα οποία λείπουν από δύο διαφορετικούς χώρους υποδοχής. Οπότε έχουμε την ίδια πληροφορία από δύο χώρους υποδοχής ή από δύο χώρες μέλη και περισσότερες. Παράδειγμα, αν ένα παιδί φτάνει, ας πούμε, στη Λέσβο, στην Ελλάδα, δηλώνεται αγνοούμενος από εκεί και δηλώνεται και αγνοούμενος και από κάποιο άλλο χώρο υποδοχής στην υπηρετική Ελλάδα και ίσως αργότερα να δηλωθεί ως αγνοούμενος από κάποια άλλη δομή υποδοχής στη Σουηδία ή οποιασδήποτε άλλη χώρας έπειτα δεν ξέρουμε πόσα από αυτά τα παιδιά βρίσκονται τελικά και πού. Κάποια από αυτά τα οποία αγνοούνται από την Ελλάδα, από την Ιταλία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, καταλήγουν σε μια άλλη χώρα μέλος, στην Αυστρία ας πούμε. Όμως οι αυστριακές αρχές δεν ξέρουν κατά πόσο το παιδί αυτό είναι αγνοούμενο και ούτε και οι ελληνικέ αρχέ γνωρίζουν ότι το παιδί αυτό έχει εμφανιστεί στην Αυστρία, έχει βρεθεί εκεί. Οπότε ο κηδεμόνας ή οποιαδήποτε άλλη υπεύθυνη αρχή που καθορίζουν όμως θα πρέπει να δηλώνουν τέτοια συμβάντα στην αστυνομία. Η έλλειψη ο θα πρεπει να τέτοιου εντοπισμού και καταγραφής έχει σαν αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα παιδιά να μην μπορούν να βρεθούν ποτέ. Δεν έχουν κυδεμόνα ή όταν υπάρχουν κηδεμόνες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους και δεν αναφέρεται η διαδικασία αυτή ξεκάθαρα στον νόμο. Κάτι το οποίο δυσκολεύει την όλη διαδικασία. Βάσει του άρθρου 32 της ε, απόφασής μας, οι αγνοούμενοι πρέπει να συμπεριλάβονται στο ΣΥΣ 2. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Γίνεται μόνο αν πιστεύουν ότι το παιδί έχει φύγει στο εξωτερικό. Το 2015 κάπου 60.000 υπόνες υπήρχαν για αγνοούμενα παιδιά σύμφωνα με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως δεν ξέρουμε πόσα από αυτά τα παιδιά ήταν ασυνόδευτα. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε τώρα. Για την περίπτωση ασυνόδευτων παιδιών πάντως που δηλώνονται ως τέτοια στην αστυνομία, δεν γίνεται παρακολούθηση γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την έρευνα είτε μια φωτογραφία του παιδιού, είτε προσωπικές πληροφορίες, είτε δακτυλικά αποτυπώματα, είτε οτιδήποτε. Πώς λοιπόν μπορούμε να βοηθήσουμε την έρευνα με στοιχεία. Πρώτα απ' όλα όλες οι περιπτώσεις αγνώμενα ασυνόδευτων παιδιών πρέπει να φτάνουν στην αστυνομία και να μπαίνουν στο ΣΥΣ 2. Έπειτα, οι κηδεμόνες πρέπει σαφώ να έχουν την υποχρέωση ότι μέσα στι 24 ώρες πρέπει να δηλώνουν ότι το παιδί είναι αγνώμενο. Έπειτα, τα συνόδευτα παιδιά θα μπορούσε για να είναι πιο ορατά, να προβληθούν περισσότερο, να καταχωρηθούν σε μια ειδική κατηγορία. Έτσι θα βοηθούσε αυτό, εφόσον βέβαια προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, να βοηθήσει στη διερεύνηση των υποθέσεών τους και να βρεθούν οι αρχέ προστασία των παιδιών θα έπρεπε έμεσα ή άμεσα να έχουν πρόσβαση στο ΣΥΣ2. Έπειτα δεν θα πρέπει να δημιουργούμε έναν φαύλο κύκλο όπου βρίσκονται τα γνώμενα παιδιά και μετά εξαφανίζονται εκ νέου. Θα πρέπει πρώτα να καταλαβαίνουμε γιατί καταχωρήθηκαν ως αγνούμενα, τι έγινε, γιατί φύγαν, που πήγαν και έτσι να αποφύγουμε την επανάληψη του φαινομένου. Η κάθε περίπτωση θα πρέπει να το χωρί χωριστά. Ξέρουμε ότι πολλά από τα ασυνόδευτα παιδιά φεύγουν από του χώρου υποδοχή προσπαθώντα να βρουν του γονεί του ή οικογένεια που έχουν σε κάποια άλλη χώρα μέλο. Ξέρουμε επίση ότι επειδή κρατούν πολλοί οι διαδικασίε και το διοικητικό άκρο είναι τεράστιο και είναι δύσκολε οι σχέσει με τι αρχέ, οδήγησαν αποτέλεσμα τα παιδιά να μην ενημερώνονται επαρκώ και να καταλήγουν να φεύγουν και να ταξιδεύουν μόνο τους, κάτι το οποίο τα καθιστά βέβαια εύκολα θύματα συμμοριών. Κανένα παιδί δεν θέλει να μείνει πίσω από σειρματόπλεγμα σε κλειστές δομές αν δεν έχει την κατάλληλη περιποίηση και δεν είναι σίγουρο ότι θα αποφύγει την κακοποίηση. Έπειτα νιώθουν ε, ότι θα απορριφθεί η αίτησή τους ε, για το άσυλο. Προσπαθούν πολλές φορές τα παιδιά από μόνα τους να ζήσουν, προσπαθώντας να βρούνε μέλη της οικογένειάς τους. Τι κάνουμε λοιπόν όταν ε, εξαφανίζεται ένα παιδί. Πρώτα απ' όλα όλοι οι παράγοντες, οι αρχές για το άσυλο, οι δικαστικές αρχές αλλά και οι αρχές προστασίας του παιδιού πρέπει να συνεργάζονται. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι αρχές τηρούν την αρχή που είναι το προτιμότερο συμφέρον για το παιδί. Να δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ασυνόδευτους, με μέρημνα, με προποθέσει τέτοιε που να τα βοηθούν να μεγαλώσουν σε προστατευμένο περιβάλλον. Και τρίτον, πρέπει φυσικά να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να φτάνουμε στους εγκληματίες και να τους διώκουμε. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι Ποτέ τα παιδιά δεν θα φύγουν από έναν χώρο στον οποίο αισθάνονται ότι προστατεύονται παρκώς και τα φροντίζει. Μόνο αν υπάρχουν τέτοιοι χώροι θα μειωθεί ο αριθμός των αγνούμενων παιδιών. Να ενισχύσουμε επίσης τις δομές υποδοχής, είτε πρόκειται για ανάδοχες οικογένειες, είτε για οτιδήποτε άλλο. Είναι καλύτερα πάντως τα παιδιά να πηγαίνουν σε μικρές οικογένειες ανάδοχες παρά να μένουν σε ιδρύματα και σε καταβλισμούς. Πάντα, πάντως, τα παιδιά πρέπει να παραμένουν στο σύστημα προστασίας των παιδιών. Και όταν μπαίνουν στη διαδικασία της εισασύλου, πάλι να εμπλέκεται σε αυτό και η υπηρεσία προστασίας των παιδιών. Τώρα, τα μέτρα όπου τα παιδιά μπαίνουν σε κάποιες ε, δομές τα παιδιά προστατεύονται γιατί αν πριν ήταν στα χέρια κάποια συμμορίας αποκόβονται από αυτήν. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να τα προστατεύουμε και να αξιολογούμε τον κίνδυνο επιστροφής τους σε τέτοιες συμμορίες και να ξέρουμε για πόσο καιρό τα κρατάμε και να αναθεωρείται η απόφαση κάθε τόσο. Είτε πρόκειται για κλειστές δομές είτε όχι, τα παιδιά δεν πρέπει να κλειδαμπαρώνονται επειδή απλώς και μόνο θεωρούν ότι έτσι τα προστατεύουν περισσότερο. Όχι, έτσι δεν βοηθάνε ούτε τα συγκεκριμένα παιδιά και σίγουρα όχι άλλα τα οποία βλέποντα αυτή την κατάσταση με τίποτα δεν θα δεχτούν να μπουν σε δομέ και θα προτιμήσουν να κυκλοφορούν ε, μόνα τους ε, χωρίς να έχουν ε, καταχωρηθεί πουθενά. Έπειτα, οι φύλακες των δομών θα πρέπει να εντοπίζουν πολύ γρήγορα τον κίνδυνο που ελοχεύει στις περιπτώσεις κάποιων παιδιών. Και τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται, ανάλογα βέβαια με την ηλικία τους. Προκειμένου πάντως να υπάρχει εμπιστοσύνη, πρέπει να τους λέμε την αλήθεια και να συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες τους και τους φόβους τους. Τέλος, για να γίνει πραγματικότητα η ενοποίηση των οικογενειών, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσπαθούμε να πετύχουμε, γιατί έτσι μειώνεται το αίσθημα της ανασφάλειας και τα παιδιά γίνονται λιγότερο ευάλωτα σε καταχρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Δημητροπούλου. Η κυρία Μοράλης ε, από τη Missing Children Europe. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, το πρόβλημα των συνόδευτων ε, ε με, ε, παιδιών μεταναστών που λείπουν ε, υπάρχει εδώ και χρόνια και όπως φαίνεται λαμβάνει νέες διαστάσεις το πρόβλημα. Η Missing Children Europe για να ανταποκριθεί σε αυτό το ζήτημα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2014 για την πρόληψη και την ε, αντιμετώπιση του προβλήματος. Το πρόβλημα συνίσταται σε έρευνα με επαγγελματίε τη επιβολή του νόμου, τα κέντρων υποδοχή ε, και των σχετικών υπηρεσιών ε, για τα ε, αγνώμενα παιδιά σε διάφορε χώρε. Τα ευρήματα δείχνουν κάποια συνοχή και επιβεβαιώνουν διάφορε προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για την προστασία τους. Η πρώτη πρόκληση είναι η έλλειψη εκπαίδευση των επαγγελματιών. Κανένας από τους εκπροσώπους των αρχών επιβολής των νόμου δεν είχε λάβει τη σχετική εκπαίδευση. Μόνο το 22% των κυδεμόνων ε, και των υπευθύνων κηδεμονίας ε, είχαν εκπαιδευτεί και ελάχιστη για την αντιμετώπιση της εξαφάνισης τέτοιων παιδιών. Πολύ συχνά οι υπευθύνοι θεωρούν ότι όταν αυτά τα παιδιά εξαφανίζονται ε, έχουν εξαφανιστεί από διαβούληση. Μια δεύτερη πρόκληση αφορά την έλλειψη διαδικασιών πρόληψης. Όταν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες εφαρμόζονται τοπικά και συχνά δεν είναι γνωστές από τους, από υπευθύνους. Η μελέτη δείχνει ότι έλλειψη εκτίμησης κινδύνου για τα παιδιά που εισέρχονται στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Η έλλειψη συνεκτικών διαδικασιών ε, δυσκολεύει την εξέβρεση των παιδιών. Οι διαδικασίες ε, ε αναφόρας ε, είναι επίσης δύσκολες. Πολύ συχνά υπάρχουν καθυστερήσεις ή οι υποθέσεις δεν αναφέρονται καν. Συνήθως ε, δεν ακολουθούνται από κάποια διαδικασία. Διάφορα δίκτυα, όπως οι τηλεφωνικές γραμμές για τα εξαφανισμένα παιδιά, που λειτουργεί σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν λειτουργεί επαρκώς Επίσης, πολύ συχνά οι περισσότεροι και δαιμόνες αναφέρουν ότι ενώ ορισμένα παιδιά έχουν βρεθεί, ε, συχνά αυτοί δεν ενημερώνονται. Η έκθεση δείχνει διάφορες προκλήσεις που υπάρχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφορών οργανισμών για τα ασυνόδευτα παιδιά ε, μετανάστες. Ε, έτσι παρεμποδίζεται η πρόληψη και η αντιμετώπιση. Επίσης ε, δεν υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία. Η ανταλλαγή πληροφοριών ε, σπάνια λαμβάνει χώρα. Επίσης αναφέρεται ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά εξαφανίζονται διότι αποθαρρύνονται από την πολυπλοκότητα των νόμιμων διαδικασιών που θα τους επέτρεπε την επανένωση με τις οικογένειές τους. Αλλά παιδιά εξαφανίζονται λόγω φόβου να σταλούν πίσω στη χώρα τους Στη Σουηδία ο βαθμός εξαφάνισης μειώθηκε όταν αναστάλησαν οι διπλές μεταφορές στην Ελλάδα, το οποίο δείχνει πόσο επηρέασαν αυτές οι μεταφορές, αυτές ε, τις εξαφανίσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Την περασμένη εβδομάδα εκδώσαμε ένα εγχειρίδιο για επαγγελματίες με οδηγίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του προβλήματος το εγχειρίδιο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας κατάρτισης για επαγγελματίες οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι ενώ το εγχειρίδιο έχει πρακτική εφαρμογή χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση και περισσότερους πόρους στη χώρα τους για να κάνουν τη δουλειά τους. Απαιτούνται προσπάθειες ώστε οι οργανισμοί να συμφωνούν σαφείς διαδικασίες και ρόλους σε εθνικό επίπεδο για βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνου, της υποβολής αναφορών και των ε, αποκρίσεων. Επίσης χρειάζονται διαδικασίες, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν οι λόγοι που οδηγούν σε εξαφανίσεις. Η οικογενειακή επανένωση πρέπει να λαμβάνει προτεραιότητα. Τα παιδιά θα πρέπει να υποβάλουν τις ασύλου στην χώρα όπου βρίσκονται χωρίς να μεταφέρονται σε άλλες χώρες. Οι κηδεμόνες πρέπει να ορίζονται άμεσα μόλις αφηχθεί το παιδί. Επίση, τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται για αυτέ τι διαδικασίε, επειδή πολύ συχνά οι μόνε προφορέ στι οποίε βασίζονται είναι αυτέ που έχουν λάβει από διακινητέ καθοδών. Τρίτον, η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να βελτιωθεί για την αντιμετώπιση αυτών των εξαφανίσεων. Αυτό θα απαιτούσε ανταλλαγή πληροφοριών των αρχών, καθώς και κοινέ ερευνητικές ομάδες που θα αναλύουν πληροφορίες και τα δίκτυα διακίνησης και θα ε, βοηθούν στην αποσάρθρωσή του. Πολλά δίκτυα όπως το ΣΥΣ και τα hotline για τα εξαφανισμένα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά. Τέλος, οι αρχέ τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ολοκληρωμένα συστήματα προστασία των παιδιών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο μια ολοκληρωμένης προσέγγιση για τα εξαφανισμένα παιδιά μετανάστες. Μία από τις αρχές αυτές της Κομισιόν είναι ότι κάθε παιδί αναγνωρίζεται και προστατεύεται ως κάτοχος δικαιωμάτων με αναμφισβήτα, αδιαμφισβήτα δικαιώματα. Μόλις εξαφανιστεί ένα παιδί, εξαφανιστεί και η προστασία. Η απόκριση στην εξαφάνιση τέτοιων παιδιών δεν πρέπει να εξαρτάται από το αν είναι υπήκοοι ή αν είναι ε, ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μοράλες πολύ σοβαρά τα ζητήματα που αναφέρατε. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Έχω επτά μέλη που επιθυμούν να λάβουν τον λόγο και ξεκινάμε τον κύριο Λένερ. Παρακαλώ. Thank you. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά αυτά που ακούσαμε. Δεν ξέρουμε για πόσα παιδιά μιλάμε, ούτε που βρίσκονται, ούτε με ποιον, τι κάνουν. Εντάξει, είναι να λέτε ότι δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, όμω δεν μπορείτε να λέτε πως δεν έχουμε καθόλου αποδεικτικά στοιχεία και ότι μπορεί να είναι στα χέρια ε, δουλεμπόρων ή ε, να δουλεύουν ως σκλάβοι εκμετα... σε... και να είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Μα ζητήσατε βοήθεια και παρατήρησα πως δύο από εσάς μίλησαν ε, σχετικά με το να ε, μειωθεί η ηλικία καταγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων ε, στο σύστημα Eurodac, να γίνεται από 14 χρονών και πάνω. Αυτό δεν ξέρω αν βοηθά την κατάσταση, δεν ξέρω αν είναι τεχνικά εφικτό, ε, διότι τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία που μεγαλώνουν ακόμα και ίσως υπάρχει πρόβλημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τώρα, σε σχέση με τους κανόνες του Δουβλίνου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν άσυλο που, όπου και αν βρίσκονται και όχι μόνο στην ε, χώρα που φτάνουν πρώτη φορά. Επίσης, πολλά παιδιά μπορούν να φοβούνται να καταγραφούν, να φοβούνται τις αρχές, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν άκουσα πολλά θετικά από μη κυβερνητικέ οργανώσει σχετικά με τη συνεργασία του με την Ευρωπόλ και είναι σημαντικό να τονιστεί αυτό. Επίση, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπόλ αν αισθάνεστε ότι μπορείτε μαζί με τι ε, ΜΚΟ, με το Missing Children ή με άλλε, ότι έχετε τι ικανότητε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν σήμερα τα αγνοούμενα παιδιά, είτε είναι αγνοούμενα από ε, τις χώρες τις οποίες αγνοούνται, είτε είναι ε, μετανάστες, πρόσφυγες, ε, ζητούν άσυλο, είναι παιδιά. Τελεία και παύλα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα, διότι κάθε δευτερόλεπτο που περνά μειώνει και τις πιθανότητες να βρεθεί ένα παιδί. Και τι κάνουμε εδώ. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι οι εθνικές αρχές δεν είναι τόσο ε, ενημερωμένες όσο πρέπει. Στη δική μου περιοχή, στη Νότια Ολλανδία, συνορεύουμε με τη Γερμανία και το Βέλγιο. Ε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα ε, ήταν δύο παιδιά αγνοούμενα από ένα κέντρο υποδοχής. Θα μπορούσαν να είναι στο Βέλγιο, στη Γερμανία, οπουδήποτε. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φεράρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να επισημάνω δύο ζητημάτα. Το πρώτο αφορά τα παιδιά κάτω των 16 που έχουμε σε κέντρα υποδοχής ε, στην Ιταλία, στην Καλαβρία, στην Καλαβρία ειδικότερα ένα πρόβλημα που έχω δει εγώ αφορά την έλλειψη εθελοντών. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε πολύ. Δεν έχουμε πολλούς τέτοιους ε, κηδεμόνες ε, εθελοντές και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, πρόβλημα σύγκρουσης συμφορέντων. Λόγω της έλλειψης τέτοιων κηδεμόνων ορίζονται κηδεμόνες ή διαχειριστές των κέντρων και αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε σύγκρουση συμφορέντων διότι τα συγκεκριμένα άτομα δεν χαρακτηρίζονται από την αμεροληψία που θα έπρεπε και που θα είχε ένας και Και μετά υπάρχει το πρόβλημα της ε, σχέσης μεταξύ κηδεμόνων και ε, ασυνοδευτών ανηλίκων πολλές φορές, και του σχετικού αριθμού. Πολλές φορές ένας κηδεμόνας είναι υπεύθυνο για 70 ασυνοδευτά ανηλικά παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να μπορεί να τα παρακολουθεί με την ε, πρέπουσα προσοχή. Είναι πολύ ψηλό ο αριθμό. Ένα άλλο πρόβλημα αφορά το σχολεία. Πολλά ε, ανήλικα παιδιά, 15, 16, 17 ετών, χρειάζονται μαθήματα ε, αλφαβητισμού ουσιαστικά που πολλές φορές δεν έχουν προβλεφθεί από το κράτος έτσι, βραδινά μαθήματα ε, επίπεδου δημοτικού σχολείου. Και έτσι λοιπόν παιδιά 5-6 ετών ε, που πηγαίνουν στο δημοτικό έχουν υψηλότερο επίπεδο από αυτά τα παιδιά των 16-17 ετών. Έτσι λοιπόν αυτά τα συνόδευτα παιδιά, επειδή δεν θέλουν να, να τα βάλουν στις ίδιες τάξεις, τα παιδιά αυτά 15-17 ετών δεν πηγαίνουν στο σχολείο και έτσι δεν μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν τη γλώσσα, να μάθουν να, αποκτούν σχέσεις με τη χώρα που βρίσκονται. Έτσι λοιπόν τα ανήλικα αυτά παιδιά ε, κυκλοφορούν ελεύθερα στις πόλεις και είναι εύκολα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ε, ή της χειραγώγησης από οποιονδήποτε τους προσφέρει κάποια δουλειά. Ε, μια άλλη ερώτηση όσον αφορά την, ε, τον οργανισμό ΦΡΑ, τον ορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, σχετίζεται με την αξιολόγηση του ενδεχόμενου ανάθεσης των ασυνόδευτων ανηλίκων σε ιδιώτες και σε οικογένειες ίσως. Πάντα τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση κάτι τέτοιο. Ε, ε, ε προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ανηλίκων ε, δεδομένης της έλλειψης εθελοντών και δαιμόνων. Ευχαριστούμε κυρία Φεράρα να ζητήσω από τους συναδέλφους να συντομεύουν διότι δεν θα προλάβουμε. Η κυρία Κορέτζα Μπίλτ παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή που έχουμε για αυτό το τρομερό ζήτημα. Ήδη στην ε, ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού αρχίσαμε τη συζήτηση μετά από την επίσκεψη της εκπροσώπου του Missing Children Europe και μα μας είπε μας εξέπληξαν. Στις πολιτικές ε, ομάδες λοιπόν αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια διακοινοβουλευτική ομάδα και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σήμερα και μπορούμε ανοιχτά να συζητήσουμε και με όλους τους συναδέρφους το ζήτημα είναι πάντα πολύ απογοητευτικό. Αυτό που λέτε εσείς είναι ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ούτε διασυνοριακά μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου, ούτε τίποτα. Οπότε έρχομαι τώρα στην καταχώρηση. Το να παίρνει κανείς δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να το θεωρήσει σαν κάτι αρνητικό, κακό για τα παιδιά γιατί ένας 14χρονος, και η Λάρα ήταν ε, αρμόδια για το άσυλο, για την εργασία που κάναμε για το άσυλο, αλλά εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι η καταχώρηση, τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι ο τρόπος που έχουμε ώστε τα παιδιά να ενταχθούν σε ένα σύστημα προστασίας. Γιατί έτσι οι αρχές γνωρίζουν ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονται στην Ευρώπη και άρα μπορούμε και να τα προστατεύσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι δυστυχώς το 50% των ε, παιδιών μεταναστών δεν φτάνουν καν στους καταβλισμούς γιατί έχουν συναντηθεί με λαθροδιακινητές και συμμορίες και έτσι δεν εντάσσονται ποτέ στο σύστημα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν περισσότερο, αναφερθήκατε στο Eurodac, το SIS1, το SIS2, διαβατήρια παιδιών. Προς το παρόν δεχόμαστε την αναγνώριση προσωπικών χαρακτηριστικών. Μήπως θέλουμε και βιομετρικά δεδομένα για τα παιδιά να έχουμε μια τέτοια βάση δεδομένων που να ενημερώνεται τακτικά. Και θέλω να ρωτήσω κάτι τη Europol. Διότι εσείς βέβαια βρίσκεστε υπό πίεση. Εσείς πρέπει μέρος των ε, πηγών σας να αφιερωθούν στην τρομοκρατία, κατά πολέμηση της τρομοκρατίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι απόλυτα θεμητό και δεν ε, σας επικρίνω γι' αυτό, απλώς ρωτάω. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να είναι σε βάρος του εξαιρετικού έργου που κάνετε για την καταπολέμηση των παιδιών που πέφτουν στα χέρια των ε, συμμοριών και λαθροδιακινητών. Ενώ μαθαίνουμε ότι πρόκειται όλο περισσότερο για παιδιά ασυνόδευτα, κορίτσια, ως επιτοπλίστων που μας φτάνουν. Είναι μαζικό το φαινόμενο. Οπότε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε αρκετούς πόρους και θα μπορείτε πραγματικά να ασχοληθείτε με την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση, όλα αυτά που τόσο καλά μας περιγράψατε δηλαδή μέχρι τώρα, προκειμένου τα παιδιά να μην πέφτουν στα χέρια συμμοριών και κλιματικών ε, ομάδων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δύο τρία λεπτά το πολύ ο καθένας παρακαλώ. Δεν μπορώ να σας ε, υποχρεώσω αλλιώς, σας το λέω. Παρακαλώ. Εσείς. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιούρεκ. Το θέμα των αγνώμενων παιδιών που συζητάμε σήμερα την Ιεμένη, την Σομαλία, τον Ταρφούρ δεν τέθηκε τίθεται εδώ στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι μια χωρίς προηγούμενο τραγωδία. Καλό θα ήταν να μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Γιατί ακόμα και αν ο αριθμός των παιδιών που έχουν βρεθεί είναι μικρός, και εδώ πολύ θα ήθελα να ξέρω πόσα παιδιά τελικά έχουν βρεθεί από τα γνώμενα, Ακόμα και από αυτό το μικρό δείγμα μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Πρέπει να ρωτήσουμε τι ακριβώς συνέβη. Είτε τα παιδιά αυτά απήχθησαν, απάγονται σε τεράστια κλίμακα ή κάπου υπάρχει απάτη. Τα παιδιά αυτά δηλαδή αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και δεν μπορεύονται κάποιοι. Ίσως οι πληροφορίες για τα παιδιά τα οποία μπήκαν στις χώρες μας να φουσκώνεται για να κρυφτούν άλλοι οι οποίοι μπαίνουν στις χώρες μας. Τα παιδιά όμως πρέπει να τα προστατεύσουμε. Η εκπρόσωπος του Missing Children το είπε. Πράγματι, όλες οι χώρες μας έχουν συνταγματικούς κανόνες που λένε ότι όλοι χαίρουν προστασίας, ότι προστατεύουμε την ακερότητα και την αξιοπρέπεια όλων. Δεν θέλω να βγάλω εύκολα συμπεράσματα ή να κατηγορήσω κανέναν, γιατί ξέρω ότι η Europol κάνει ό,τι μπορεί. Έχετε περιορισμένους πόρους κι εσείς. την κύρια ευθύνη την έχουν υπηρεσίε επιβολής του νόμου των χωρών από όπου εξαφανίζονται τα παιδιά. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα επίσης έχουν ευθύνη, γιατί έχουν αγνοήσει τη δυνατότητα αυτή. Λένε να ανοίξουμε τις πόρτες μας σε όλους, χωρίς να καθίσουν και να σκεφτούν τα ζητήματα της ασφάλειας που απορρέουν. Διότι, επαναλαμβάνω, ή που έχουμε να κάνουμε με εγκληματικές ενέργειες σε μια τεράστια κλίμακα ή αλλιώς υπάρχει τεράστια έλλειψη ευθύνη από πλευρά των θεσμικών οργάνων και από τι κυβερνήσει των χωρών μελών που έχουν ενθαρρύνει του μετανάστε να έρθουν στι χώρε μα. Και τα ασνόδευτα αυτά παιδιά πληρώνουν την ύφη. Γιατί στι περισσότερε περιπτώσει τα παιδιά δεν έχουν έρθει με τη θέλησή του, τα φέραν εδώ. Και συγχρόνως ακούμε ότι αυτοί που ήταν ρεαλιστές για την όλη εξέλιξη είχαν κάνει λάθος. Όχι. Αυτοί που είναι πολιτικά υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φυσικά ζούμε σε μια δημοκρατική κοινότητα όπου η δημοκρατική ευθύνη πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή. Κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Την 1η Απριλίου πήγα στη Μόρια και είδα τα παιδιά εκεί. Από τις 20 Μαρτίου και έπειτα, μετά τη συμφωνία δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, μόνο 2.500 άνθρωποι έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ στη Μόρια είδα παιδιά υποκράτηση και ξέρω ότι είναι ακόμα περισσότερα από αυτά που είδα. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, είναι όμως γεγονός. Και είδα παιδιά στα αυτοσχέδι, στους αυτοσχέδιους καταβλισμούς στον Πειραιά, αλλού στην Ελλάδα, είδα παιδιά στην Ιδωμένη, πολλά από αυτά συνόδευτα ή με ανθρώπους που έλεγαν πως είναι συγγενείς τους ή με διάφορους ε, χωρικούς. Ήμουν στη Λέσβο, σε ένα σπίτι που μία ΜΚΟ, συνεργαζόμενη με τις ελληνικές αρχές, ε, σύτιζε 7 ανήλικους. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν μόλις 7 χρονών και μας είπαν ότι δεν έχουν αρκετές εγκαταστάσεις, δεν έχουν αρκετούς ε, δασκάλους, δεν έχουν αρκετούς ε, που θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτά τα παιδιά. Πολλά από αυτά τα παιδιά βρίσκονται εκεί θύματα των διακινητών θύματα ε, κάθε είδους απεχθών εγκληματικών οργανώσεων. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Συμβαίνει στην Ευρώπη και είναι απαράδεκτο. Και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για αυτό το χάλι στην Ευρώπη. Πολλά ε, από αυτά τα παιδιά είχαν μητέρες που, που τα περίμεναν περίμεναν να επανενωθούν οι οικογένειες, είχαν πατέρες, ε, συγγενείς που περίμεναν στη Γερμανία, στη Σουηδία την οικογένειά τους, τα παιδιά τους και πολλά από αυτά ταξίδεψαν μόνα ακριβώς γιατί δεν υπήρχε, ε, ακριβώς γιατί περίμεναν να επανενωθούν και κάποια κρατημέλη αποφάσισαν να καταστρέψουν το Σέγγεν και να κλείσουν τα σύνορα. Γι' αυτό πράγματι, αν δεν δείξω με το δάχτυλό μου την Ευρωπόλ και τις άλλες υπηρεσίες που προσπαθούν να κάνουν κάτι, θα το κάνω και θα δείξω τις κυβερνήσεις μας, οι οποίες έχουν την πολιτική ευθύνη και έχουν αποτύχει στα καθήκοντά τους, το καθήκον τους να προστατεύσουν αυτά τα παιδιά, τους πρόσφυγες, ε, τα παιδιά μετανάστες, Και το μόνο που κάνουν μετά από αυτή τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση και Τουρκία είναι να αφήσουν αυτά τα παιδιά να γίνουν ε, λία εγκληματιών. Δεν έχουν αναλάβει τι πολιτικές τους ευθύνε. και έχουμε τα κράτη-μέλη στην πρώτη γραμμή που παραβιάζουν το χώρο του Σέγγεν, έχουν μπλοκάρει τα σύνορα και ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό. Συμπεριλαμβάνεται και η Γερμανία σε αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίνμπεργκ έχει το λόγο. Συγγνώμη. Η Γερμανία στην αρχή μας έλεγε δεν υπάρχουν σύνορα και μετά στην ουσία βοηθούσε τους άλλους να τα κλείσουν. Συγγνώμη, έχουμε έξι άτομα που ζητούν το λόγο, λέει η Πρόεδρος, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Κυρία Βίνμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Καταρχάς θα ήθελα να πω πως είναι ανησυχητικό αυτό που διαβάζουμε, ότι αυτά τα παιδιά γίνονται σεξουαλικοί σκλάβοι, πέφτουν θύματα εγκληματικών οργανώσεων. Σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι, διότι δεν επιτρέπεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι με τη μαζική μετανάστευση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι περίεργο να βλέπουμε παιδιά να ταξιδεύουν μόνα τους. Πέρυσι πάρα πολλές χιλιάδες παιδιά συνόδευτα έφτασαν στη Σουηδία και εξαφανίστηκαν, αγνοούνται. Πιστεύω πως ε, τώρα έχει προκύψει ένα νέο πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνδρες που έρχονται από το Αφγανιστάν και από άλλες χώρες και ζητούν άσυλο ε, τους αρνείται το άσυλο. Τι γίνεται με αυτούς. Ξέρουν πώς θα τους απελάσουν και εξαφανίζονται. εμένα, ξέρετε πόσα ε, αγόρια από το Μαρόκο είναι εξαφανισμένα και γυρίζουν στους δρόμους της Σουηδίας. Γιατί ξέρουν πώς θα τους στείλουν πίσω στο Μαρόκο και δεν θέλουν να επιστρέψουν. Στη Σουηδία αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για το αν θα πρέπει αυτά τα παιδιά να ε, συλληφθούν, να κρατηθούν. Το πρόβλημα όμως αυτό σίγουρα δεν υπάρχει μόνο στη Σουηδία. Πρέπει να έχει απαντηθεί και σε άλλες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι αυτό. Τι τους κάνουμε όταν δεν μπορούμε να τους διώξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Λάμπερτ. Κάποιοι... Πολλοί από εμά εδώ και χρόνια λένε ότι αυτό το σύστημα που έχουμε θα πρέπει να εξετάζει και τις συνέπειες ε, για όσους δεν μπορούν να γυρίσουν στις αρχικές τους χώρες λόγω συνθήκων εκεί. Ε, σε πολλά κράτη-μέρη λοιπόν υπάρχει κίνδυνος να τιμωρούμε παιδιά λόγω της ανευθυνότητας, λόγω των χρόνων καταγωγής τους, ε, στις χώρες καταγωγής τους ή στα δικά μας συστήματα. Και τώρα βλέπουμε αυτές τις προτάσεις για να αλλάξουμε το σύστημα ασύλου. Και εγώ ανησυχώ, διότι ένα από τα πράγματα που συμπεριλάβαμε σε αυτές τις ε, αναδιατυπώσεις ε, ήταν ε, η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των παιδιών και τα όσα ακούσαμε σήμερα μας δίνει πολύ καλές ενδείξεις και οι προτάσεις, για τις προτάσεις πολιτικής που χρειαζόμαστε. Ένα από τα πράγματα που χρειαζόμαστε, πιστεύω, είναι μεγαλύτερες προσπάθειες με τις δικές μας κυβερνήσει, για υλοποίηση τη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη μη επιστροφή των παιδιών υπό το Δουβλίνο 2 ε, στη χώρα όπου πρώτα έκαναν ε, αίτηση ασύλου ε, και να δεχόμαστε την αίτηση εκεί που βρίσκονται. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, για να βελτιώσουμε τα ζητήματα καταγραφής πρέπει να βελτιώσουμε τα ζητήματα εμπιστοσύνης στο σύστημα και αυτή η εμπιστοσύνη λείπει. Ε, όταν κοιτάμε τι κάνουν οι κυβερνήσεις μας, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, όλο το θέμα του Καλέ, όπου έχουμε αποφάσεις δικαστικές που καθιστούν απόλυτα σαφέ ότι τα παιδιά στα, ε, ε, στο Καλέ έχουν δικαιώματα δυνάμει του Δουβλίνου 2 και τη συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως η νομοθεσία αυτή δεν υλοποιείται και νομίζω οι γαλλικές αρχές επίσης υπολείπονται πραγματικά στην παρακολούθηση και στην υποστήριξη των νέων αυτών ανθρώπων. Εμείς ως Κοινοβούλιο ξέρουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε και θέλω να ευχαριστήσω τους απόψινούς ομιλητές που τα παρουσίασαν τόσο καθαρά ώστε να αρχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας εμείς μαζί με τις κυβερνήσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτς, κυρία Βεζία παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, σύγχυση δι, διαβλέπω εγώ. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω από πού βρήκαμε αυτό, το 10.000, από πού βγήκε αυτός ο αριθμός και τι εκπροσωπεί. Κατάλαβα πολύ καλά ότι ο αριθμός των καταγραφών είχε αυξηθεί, ε, μιλάμε για τα παιδιά που έχουν φτάσει στην Ευρώπη, ε, αυξήθηκε αυτός ο αριθμός και τα κράτη δεν έχουν αρκετά μέσα για την καταγραφή, αλλά αυτό εμένα δεν μου εξηγεί τα πράγματα. Ούτε όταν λέμε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά πέφτουν θύματα ε, ε, λαθρεμπορίου. Υπάρχει μία τεράστια ευθύνη των κρατών. Ε, όλα αυτά τα κράτη έχουν προσυπογράψει την, το Διεθνή Χάρτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Θα πρέπει να τηρούν και το Δουβλίνο, όχι μόνο το άρθρο 1 όχι μόνο το άρθρο που επιτρέπει την επιστροφή, αλλά και αυτό που εμποδίζει την ε, ε, ε, επαναπρόθεση των ανηλικών παιδιών, τα οποία προστατεύονται, πρέπει να προστατεύονται ανεξάρτητα καθεστώτος ή ηλικίας και πρέπει να θεωρούνται παιδιά πρώτα απ' όλα. Αυτό νοούμε όταν λέμε για τα συμφέροντα των παιδιών. Δυστυχώς φοβάμαι ότι ζω σε μια χώρα η οποία δεν φαίνεται να δεσμεύεται ιδιαίτερα από αυτή τη συνθήκη. Σύμφωνα με κάποιε πρώτε προφορίε, κάθε χρόνο 10.000 παιδιά χρειάζονται προστασία. Τα μισά από αυτά ε, βλέπουν να απορρίπτονται οι αιτήσει του. Γιατί, διότι σε αυτά τα παιδιά κάνουμε ε, κάτι που ονομάζουμε δοκιμές ε, ε, αμφισβητούμενη ποιότητα και που παρεμποδίζουν ε, την προστασία ενό συγκεκριμένου αριθμού ανηλίκων. Ας ε, επιστρέψουμε σε αυτή την υπόθεση του Καλέ, πολύ σωστά το υπογραμμίσαμε. 300 παιδιά ανήλικα μόνο τους βρίσκονται στο Καλέ και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο παίζουν πινκ-πονγκ με την υπόθεση αυτών των παιδιών. Θα έπρεπε να τα αναλάβει η Γαλλία και η γαλλική κυβέρνηση θα έπρεπε να πιέσει τη βρετανική κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτή την κατάσταση, διότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά έχουν δικαίωμα οικογενειακή επανένωση στην Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειαζόμαστε λοιπόν την ανταλλαγή πληροφοριών και όπω συζητήσαμε σήμερα το πρωί, βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι καθαρά θέμα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν ώστε όλα τα συστήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κυρίως των δικαιωμάτων των παιδιών. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να δοθεί πραγματικά προσοχή να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν την επίλυση αυτών των καταστάσεων γιατί δεν μπορούμε να λέμε απλά αν ναι, 10.000 παιδιά έχουν εξαφανιστεί στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και να αναρωτιόμαστε τι εκπροσωπεί αυτό στην πραγματικότητα χωρίς να λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα αυτό όσο και τα υπόλοιπα προβλήματα που εξετάζουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βέζια. Κυρία Βόλτμανς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές. Είναι μια φρικτή η υπόθεση αυτή, τόσες χιλιάδες παιδιά να είναι αγνοούμενοι. Έχω πάει στην ε, Europol, έχω ακούσει εκεί το Missing Children και το Child Focus, έχω έρθει σε επαφή και πρέπει να πω, συνάδελφοι, ότι εμείς όταν στη γειτονιά μας ε, χάνεται ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, δεν λέω ότι συγκρίνω τα γατάκια τα σκυλάκια με τα παιδιά, αλλά μέσω στα facebook, φωτογραφίες βλέπουμε κτλ. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά συζητάει τα κατεπήγοντα για παραβιάσεις που γίνονται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Δεν είναι αυτό επίγον να δούμε τι κάνει η Ευρώπη. Έμαθα πολλά για την πρόληψη σήμερα. Συνειδητοποίηση πρώτα απ' όλα των κινδύνων. Αυτό είναι το πρώτο. Οι πολίτες δηλαδή να είναι σε γρήγορση και να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να ενημερώνονται οι αρχές αμέσως μόλις εντοπιστεί κάτι περίεργο. Τα ακούμε αυτό πολύ συχνά, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται στην πράξη. Για την τροπολογία Βίλκστρομ επίσης, που λέει ότι τα παιδιά να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άσυλο εκεί όπου βρίσκονται. Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα, είναι θύματα. Ζητάω λοιπόν από την Επίτροπο Γέροβα να φροντίσει για ένα πρόγραμμα δράσης για τους ανήλικες. Από το 2014 το περιμένουμε, είμαστε 2016 κυρία Πρόεδρε. Η Επίτροπος λοιπόν ε, θα έπρεπε να βιαστεί λίγο, να προχωρήσει και να μας παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσης. Τώρα, τρία θέματα θέλω να θίξω. Ένα για σας, κυρία Πρόεδρε. Εντάξει, εγώ είμαι εδώ αναπληρώτρια στη Λίμπε, στην ΑΦΕΤ είμαι κανονικά, αλλά οι επιτροπές μας ίσως μαζί θα έπρεπε να φροντίσουν για ένα πρόγραμμα δράσης με όλα τα στοιχεία, με όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να υπάρχει ένας έλεγχος είναι το δεύτερο. Και το τρίτο, άκουσα πολλά για την πρόληψη, τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, πώς να μειωθεί το φαινόμενο. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τα 10.000 αγνοούμενα παιδιά. Πού να βρίσκονται άραγε αυτά, στην πορνεία. Μπορούμε ακόμα να τα σώσουμε. Ε, τα σκοτώνουν για να τους πάρουν τα όργανα. Ξέρω Έχω αποβάλει και γραπτή ερώτηση πριν από δύο μήνες με 40 υπογραφές και, πάνω, και παραπάνω, αλλά δεν ακόμα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι πρόγραμμα δράσης εμείς στην Ευρώπη πρέπει να αναλάβουμε τώρα, αύριο, ώστε τα παιδιά αυτά να τα βρούμε ζωντανά. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να τα βρούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά τη μεταχείριση των παιδιών στους χώρους που ανέφερε η συνάδελφος Άννα Γκόμες, έχω δύο ερωτήσεις. Ε, εντυπωσιακή έλλειψη τροφίμων για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των νεογέννητων. Να σας δώσω έναν αριθμό στοιχείο σε παιδιά 7 ετών ε, παρέχονται 100 μιλιλίτρα ε, γάλακτος την ημέρα μόνο. Τώρα η Ευρώπη ε, της αρέσουν οι εφημισμοί ε, να χρησιμοποιούν άλλα λόγια για άλλες καταστάσεις και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε να, να θεωρήσουμε ότι αυτή η ελληπής παροχή τροφής σε ένα νεογέννητο είναι μια μορφή ε, βασανιστηρίου. Η δεύτερη μου ερώτηση, πολλά ε, ανήλικα παιδιά κοντά στα 18 αλλά όχι ακόμα 18 λένε ότι είναι ενήλικοι όταν τους ρωτάνε ώστε να μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα και να αποφύγουν την κράτηση. Και εξαφανίζεται και για αυτό το λόγο. Είναι σημαντικό αυτό που είπε μία από εσάς για το γεγονός ότι ένα παιδί πρέπει να είναι κάτοχος δικαιωμάτων, πρέπει να κατέχει δικαιώματα, διότι αλλιώς ε, παρατηρούνται αυτές οι προσπάθειες να αποδείξει κάποιος ότι δεν είναι ανήλικος ώστε να αποφύγει να καταλήξει σε κράτηση, σε κάποιον καταβλισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη. Να στραφώ τώρα στους ομιλητές μας. Έχετε πολλές ερωτήσεις. Να σας ζητήσω να είστε σύντομοι. Προσπαθήστε να απαντήσετε σε δύο με τρία λεπτά, αν είναι δυνατόν, ο καθένας σας. Λοιπόν, πρώτος ο κύριος Νόιντον. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και που με επιτρέπετε να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έχω την χρυσή λύση για όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά πιστεύω να ε, συνεισφέρουμε έστω και λίγο. Ε, εμείς έχουμε όλων των ειδών ε, τους ε, υπαλλήλους. Καταρχάς, πιστεύω πως ε, πρέπει να δημιουργηθεί μια σωστή ευρωπαϊκή διοίκηση. Χρειάζονται σαφείς αρμοδιότητες, σωστή επικοινωνία, ξεκάθαρες απλές διαδικασίες και αυτό φυσικά μας οδηγεί και στο θέμα των πόρων. Εγώ δεν θα έλεγα πώς είναι τόσο ζωφερά τα πράγματα, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα. Η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη στην περίπτωση εμπορίας ανθρώπων μας έχει δείξει ότι το 2009 είχαμε ε, θετικά αποτελέσματα. Είχαν αυξηθεί βέβαια οι περιπτώσεις ε, στις οποίες ε, κληθήκαμε να βοηθήσουμε, όμως πιστεύω πως δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση. 500 τέτοιέ περιπτώσεις είχαμε συναντήσει το 2015. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη λειτουργεί. Επίσης, έγινε λόγος για διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριών στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια τεράστια πρόοδο σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Σήμερα έχει αρχίσει ο διάλογος. Και ρωτήθηκα κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσω να απαντήσω, το αν δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αρκετά γενναιόδωρο πρόσφατα ενέκρινε μία ε, απόφαση να αυξηθούν τα κονδύλια της Ευρωπόλ. Αλλά φυσικά είναι γεγονός ότι οι πόροι μας είναι περιορισμένοι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν έχουμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, να είμαστε στα ε, ελληνικά νησιά για να κάνουμε ε, δεύτερους ελέγχους ασφάλειας, οι πόροι δεν αρκούν. Και πολύ φοβάμαι ότι με αυτόν τον ε, τόσο υψηλό αριθμό ε, αγνοούμενων παιδιών θα είναι πολύ πιθανό οι πρώτες περιπτώσεις ασυνόδευτων ανήλικων που ε, έπεσαν θύματα διακίνησης να φτάσουν στα χέρια μας. Αργότερα, ο συντονισμός και η δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε είναι τεράστιων διαστάσεων. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν έχω την χρυσή λύση. Ό,τι λέω σίγουρα δεν είναι πανάκια, όμως προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημητροπούλου, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη. Πολλέ από τις συστάσεις που ακούσαμε σήμερα ανέφεραν ε, την νομική υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη. Πρέπει να σεβαστούν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχει σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει νομοθεσία για το άσυλο, ε, για τη στέγαση των ασυνόδευτων ανήλικων σε μικρέ οικογενειακές μονάδε, για τι συνθήκε υποδοχή για του ε, κυδεμόνε των παιδιών αυτών. Υπάρχει στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Το θέμα είναι γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί οι νόμοι. Πολλά από αυτά που ακούσαμε σήμερα δεν τα ακούμε για πρώτη φορά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους. Επίσης, πρέπει να διασφαλίσουμε το συμφέρον του παιδιού. Πρέπει αυτό να είναι το κύριο μέλημά μας στην ε, ε, δημιουργία νέας νομοθεσίας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πως οι αποφάσεις δεν θα παραβλέπουν το συμφέρον και, και το μέλλον των παιδιών. Ιδιαίτερα ε, τα μικρά παιδιά. Σε πολλές περιπτώσεις, πράγματι θα είναι προς το συμφέρον του παιδιού να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα γιατί έτσι θα μπορούμε να το εντοπίσουμε. Εδώ φυσικά πρέπει να εξετάσουμε και θέματα προστασίας δεδομένων και τις ε, διάφορες ε, ασφαλιστικές δικλείδες που πρέπει να υπάρχουν έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι γίνεται θα γίνεται πάντα για το συμφέρον του παιδιού. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι άσπρο ή μαύρο, υπάρχουν και αποχρώσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Τώρα όσον αφορά την κυδαιμονία των ε, παιδιών και εδώ υπάρχουν προκλήσεις στο σύστημα. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις στην Ιταλία, στην Ελλάδα και σε αλλα κρατημέλη και υπάρχει ένα εγχειρίδιο, όπως είπα και νωρίτερα, σχετικά με την κυδομονία. Έχουμε στη διάθεση μας διάφορα εργαλεία, έχουμε συστάσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από πολλούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, υπάρχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι Missing Children, αλλά πρέπει να πιέσουμε και τα κρατημέλη να αλλάξουν την κατάσταση στο έδαφος τους, στην επικράτειά τους. Επίσης, Ας μην ξεχνάμε ότι τα αγνοούμενα παιδιά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν επηρεάζει μόνο ένα κράτος μέλος. Πολλές φορές, αν κοιτάξει κανείς τα διαθέσιμα δεδομένα, θα δούμε ότι το θέμα αυτό δεν αφορά δυστυχώς μόνο την Ελλάδα ή μόνο την Ιταλία ή μόνο το τάδε κράτος, αλλά Αυτέ οι περιπτώσει αφορούν όλα τα κρατη Πηγαίνουν από νότο προς βορρά και από ανατολή προς δύση. Όλα λοιπόν τα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσει. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε το θέμα τη διεθνού ε, διακρατική συνεργασία και αυτό μπορούμε να το κάνουμε εξετάζοντας τις ε, δυνατότητες που έχουμε να βελτιώσουμε τα εφιστάμενα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας και να συμπεριληφθούν και οι αρχές ε, επιβολής νόμου στην προσπάθεια αυτή. Επίσης, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τα διάφορα συστήματα, το Eurodactosis, και να δούμε το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν αγνοούμενους ανήλικους, για παράδειγμα. Ποιο είναι το καλύτερο σύστημα για να γίνει αυτό. Να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε να ε, γίνει πιο εύκολη η συνεργασία ανάμεσα στις αρχές. Ελπίζω Λοιπόν, όταν θα ε, επανέλθουμε με αυτό, να βοηθήσουμε σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μοράλες. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που οι ευρωβουλευτές ε, θέλουν να δώσουν προτεραιότητα. Άκουσα τις λέξεις επίγον, άκουσα τις λέξεις τώρα και πρέπει να φροντίσουμε ε, να μην μείνουμε με τη γνώση ότι λείπουν 10.000 παιδιά, αλλά να κάνουμε κάτι και για την πρόληψη. Τέθηκε το ερώτημα του ποιος είναι υπεύθυνο. Θεωρώ ότι είναι διπλή υπευθυνότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια έκθεση για τα εξαφανισμένα παιδιά, τα γνώμενα παιδιά και εκεί αναφέρθηκε ότι μόνο τέσσερα κράτη-μέλη είχαν νομικές διαδικασίες ε, για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ασυνόδευτων εξαφανισμένων παιδιών μεταναστών. Συνήθως στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχει μια περίοδος μη αντίδρασης, ενώ ξέρουμε ότι αυτή η άμεση αντίδραση είναι απαραίτητη. Σε άλλα απόκριση είναι ότι ε, μπαίνει στην άκρη το αίτημα ασύλου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ξαναδούμε το θέμα ε, βάζοντα στο επίκεντρο τα καλύτερα συμφέροντα των παιδιών, όπω λέμε, διότι είναι διασυνοριακό το πρόβλημα και το να αντιμετωπίζουμε μόνο εθνικά δεν αρκεί. Πολλέ ερωτήσει ακούσαμε και πολλά σχόλια πολύ σημαντικά που θα μα οδηγήσουν προ το μέλλον. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να δείχνουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά, να τα ακούμε για να μαθαίνουμε τις ανάγκες τους και να καταλαβαίνουμε τι απειλές αντιμετωπίζουν το καθένα. Αυτό απαιτεί κόσμο, προσωπικό, εκπαίδευση και πόρους. Επίσης απαιτεί ενημέρωση των παιδιών. Τα παιδιά δηλαδή να χειραφετούνται, να μπορούν να λάβουν αποφάσεις γνωρίζοντας τους κινδύνους, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν διαδικασίες μέρημνας προς αυτά. Επίσης απαιτεί στέγαση και η κράτηση σίγουρα δεν αποτελεί σωστή απόκριση. Φυσικά, σε πολλές χώρες αυτό αποτελεί πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πράγματι δραματική. Η απόκριση σε τέτοιες καταστάσεις ε, θα προερθεί από πολλούς τομείς και πρέπει να βασίζεται στις αρχές προστασίας των παιδιών πρώτα απ' όλα. Το ζήτημα της ένταξης ε, και σχετιστεί με το ζήτημα της εκπαίδευσης, της παιδείας όπως ακούσαμε, αυτά πρέπει να λάβουν προτεραιότητα, διότι πολλά από τα παιδιά που εξαφανίζονται ξαφνικά έχουν βρεθεί σε μια κατάσταση άνευ Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί στα μελλοντικά μας προγράμματα απόκριση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ για να μας ενημερώσετε για το φλέγον αυτό ζήτημα. πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Να περάσω μέσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ευχαριστώντας σας για την παρουσία σας εδώ. Είναι σχετικό, αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Βαλερό παρουσιάστηκε στη ΛΥΜΠΕ στις 16 Μαρτίου. Η ΛΥΜΠΕ θα εκδώσει γνωμοδότηση ω συνδεδεμένη επιτροπή υπό τον κανόνα 54, υπό το άρθρο 54. Έχουν γίνει διάφορες τροπολογίες και τώρα θα γίνει ανταλλαγή ε, απόψεων με την εισηγήτρια και τους συνεισηγητές. Κυρία Βαλέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές για την ε, εξαίρετη συνεργασία. Είχαμε πολλές ε, συναντήσεις νωρίτερα. Πιστεύω πως τώρα έχουμε καταφέρει να συμβιβαστούμε στις 95 τροπολογίες. Φυσικά και δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες, αλλά πιστεύω πως κάναμε ό,τι μπορούσαμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην ψηφοφορία. Ε, το θέμα, το πρόβλημα μάλλον εδώ δεν είναι ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Αντίθετα, οι απόψεις μας συγκλίνουν. Είναι, όπως είπε η Πρόεδρος, ότι εδώ πρόκειται για εμπορία ανθρώπων και τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα. Ε, δηλαδή υπάρχουν πολλοί τομείς οι οποίοι σχετίζονται με αυτό, αστυνομική συνεργασία, κατάρτιση ε, των αρχών, υπάρχουν οικονομικές πτυχές του προβλήματος και επίσης υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην εμπορία ανθρώπων και τη διακίνηση ανθρώπων. Προστασία των θυμάτων, προστασία των μαρτύρων, προστασία των παιδιών, ε, συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών, ευαισθητοποίηση, πρόληψη. Οι διαφορές μας, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι μεγάλες. Όπως σας είπα, συγκλίνουν οι απόψεις μας και έχουμε μικροδιαφορές σε συγκεκριμένα σημεία. Πιστεύω πως σε γενικές γραμμές η συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές ήταν πάρα πολύ καλή και η γνωμοδότηση που θα ψηφίσουμε θα είναι πολύ καλή. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε πού αρχίζουν εξωτερικές σχέσεις και πού σταματούν. Όμως, στην Επιτροπή Γυναικών και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει συζητηθεί το θέμα και εδώ θα μπορούσαμε, πιστεύω, να συνεισφέρουμε επικοδομητικά με τις ερωτήσεις μας, με τα σχόλιά μας. Αυτά από μένα. Θα αφήσω τώρα τους κοιόδες ηγητές να πάρουν το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Βαλέρο. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Σίπελ και η κυρία Κόμες. Παρακαλώ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάω εκ μέρους της Κιόδος εισηγήτριας της Κριστίν Πολκαφάκη, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα το απόγευμα. Διαβάζω λοιπόν τις παρατηρήσεις της. 95 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί με κάνουν θέλω να επικεντρωθώ στα σημεία της δικιάς μου πολιτικής ομάδας και ευχαριστώ βέβαια την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Και το θέμα της προστασίας των θυμάτων είναι σημαντικό για μας να ζητήσουμε αναθεώρηση της οδηγίας για τις άδειες παραμονής. Τα θύματα πρέπει να μπορούν να παίρνουν άδεια παραμονής, ακόμα και αν δεν είναι σε θέση να συνεργαστούν με τις αρχές. Χρειάζονται τη βοήθειά μας, την αρρωγή μας και επιπλέον πρέπει να θυμηθούμε ότι τα θύματα δεν είναι υπεύθυνα για εγκληματικές ενέργειες στις οποίες τους ανάγκασαν να συμμετάσχουν, κυρίως όταν πρόκειται για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κατανακαστική εργασία. Όσον αφορά τα συνόδευτα παιδιά, πρέπει να υπάρξει μία ταυτοποίηση των παιδιών που είναι θύματα. Πρέπει να υπάρξουν κυδεμόνες για όλα τα συνόδευτα παιδιά. Εδώ πρόκειται για την εμπορία ανθρώπων, αλλά πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην εμπορία ανθρώπων και την λαθροδιακίνηση των μεταναστών. Ακόμα και αν συνδέονται τα δύο φαινόμενα, υπάρχει διάκριση. Γιατί στη μία περίπτωση το θύμα κατά κάποιο τρόπο δίνει τη συγκατάθεσή του. Η αστυνομία λοιπόν και οι δικαστικές αρχές πρέπει να καταπολεμήσουν την ε, εμπορία ανθρώπων. Από την άλλη μεριά οι ακτοφύλακες πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Να αναγνωρίζεται επίσης το καθεστώς των θυμάτων. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα δομή για την προστασία των ε, θυμάτων, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προθυμία. Αυτό όμω είναι που θέλω να τονίσω και εγώ με την τροπολογία μου 51. Τέλος, επιμένω στην αναγκαιότητα να υπάρχει αρμοδιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να υπάρξει πλήρης αμοιβαία αναγνώριση όταν πρόκειται για μέτρα προστασίας θυμάτων εμπορίες ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει εγγύηση από τις δικαστικές αρχές μιας χώρας. Η αρμοδιότητα αυτή δεν πρέπει να δοθεί σε μια νέα δομή, αλλά σε μια ήδη υπάρχουσα ευρωπαϊκή υπηρεσία. Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να δέχονται βοήθεια, να αναγνωρίζεται το καθεστώ τους όταν ταξιδεύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα ενισχυθεί η αναγνώριση του καθεστώτος του θύματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χουλμάγερ. Καταρχάς πιστεύω ότι τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων χρειάζονται προστασία. Είναι αυτονόητο. Ε, Α μην συγχαίουμε τα πράγματα. Τι σημαίνει προστασία. Προστασία σημαίνει ότι το θύμα, το θύμα βιασμού, το θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, το θύμα ε, σεξουαλικής κακοποίησης ε, χρειάζεται και οφείλει να λαμβάνει τη βοήθειά μας. Υπάρχουν επίσης και οι περιπτώσεις ανθρώπων που δουλεύουν στη μαύρη αγορά. Αυτό ε, δεν ε, σημαίνει πως έχουν την ίδια ανάγκη για βοήθεια με ένα θύμα βιασμού. Για παράδειγμα, πρέπει να κάνουμε μια, ε, έναν διαχωρισμό και να δώσουμε την πλήρη στήριξή μας στα θύματα, αλλά από την άλλη, εκείνοι που από μόνοι τους εξαφανίζονται, δεν πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Μετά αναφέρθηκε ότι υπάρχει απροθυμία από ορισμένα κράτη-μέλη να ε, βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή. Εδώ πρέπει να ζητήσουμε τη συνδρομή της Frontex έτσι ώστε να χτυπήσουμε στοχευμένα εκείνους που εκμεταλλεύονται ε, την, την ε, μεταναστευτική ε, και η προσφυγική ροή. Πρέπει να γίνει, σας είπα, ο διαχωρισμός, διότι είναι όπως ε, ακριβώς γίνεται ένα αλκοτέστ, ας πούμε. Δεν θέλεις να πιάσεις κάποιον που ήπια ένα από το, αλλά αυτόν που ήπια παραπάνω από το όριο. Η εφορία δεν κυνηγάει αυτόν που ξέχασε από προσεξία ή χωρίς να φταίει να βάλει κάτι στη δήλωσή του, αλλά εκείνον που εσκεμμένα εξαπατά το κράτος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ε, σε αυτού, ανάμεσα σε ε, αυτούς που εκμεταλλεύονται και στα θύματα. Γι' αυτό χρειάζεται και η βοήθεια της Frontex έτσι ώστε να εντοπίσουμε αυτούς που εκμεταλλεύονται τις ε, προσφυγικές ροές και παράλληλα, τιμωρώντας τους ενόχους, να βοηθήσουμε και τους πρόσφυγες, οι οποίοι χρήζουν προστασίας. Και να αποφύγουμε αυτοί οι άνθρωποι να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χολμάιρ. Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως είπατε και αυτό έχει σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Και είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε τα θύματα, αλλά και να δούμε ποιοι έρχονται ήδη ω θύματα ή ποιοι έρχονται και μετά γίνονται θύματα, διότι η κατάσταση που βρίσκονται είναι πολύ ευάλωτη. Εγώ είδα ότι στον Πειραιά κανείς δεν νοιάζεται, κανείς δεν πάει σε αυτούς τους ανθρώπους, κανείς δεν τους βοηθά να καταπολεμήσουν αυτούς τους ε, λαθρέμπορους και κανείς δεν βοηθά τις γυναίκες και τα παιδιά εκεί. Και όπως είπε και η συνάδελφος, πρέπει να αναγνωριστεί ε, το καθεστώς ε, του θύματος. Αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι όλα μπλοκαρισμένα. Δεν λειτουργεί ε, τίποτα. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν γυναικόπαιδα που περιμένουν να ενωθούν με τους συγγενείς τους σε άλλες χώρες και δεν ξέρουν πώς να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση, διότι δεν τους βοηθά κανείς. Κανείς δεν τους ε, πλησιάζει και οι προσπάθειές μας δεν έχουν αποτέλεσμα. Είναι τα πάντα μπλοκαρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, εάν παραδεχτούμε και αναγνωρίσουμε την ιδιότητα του θύματος, ε, αυτό θα βοηθήσει. Α, και πρέπει να μπει στις προτεραιότητές μας. Και πώς συνδέεται αυτό με την προηγούμενη συζήτηση. Δεν αρκεί μόνο το να ακούμε τους εμπειρογνώμονες. Πρέπει να φέρουμε εδώ το Συμβούλιο που θα μιλήσει εκ μέρους των κυβερνήσεών μας και να μας ε, πει τι γίνεται, τι κάνουν. Ελληνικέ αρχές δεν μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα διότι δεν διαθέτουν τα μέσα για να το κάνουν. Τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευση, εμπορία. Τι γίνεται για να αντιμετωπιστούν αυτά τα δίκτυα των διακινητών. Ε, πήγα πρόσφατα στην Κύπρο και στο βόρειο τμήμα και είδα πάρα πολλούς Νιγηριανούς γυναίκες οι οποίες ήταν θύματα ε, κυκλωμάτων πορνείας ε, από τον τουρκικό στρατό που τους διοχέτευαν μέσω της ε, Βόρειας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιαφέρεται κανείς για αυτά. Ενδιαφέρεται κανείς για την καταπολέμηση αυτών των κυκλωμάτων στην Τουρκία και στη Βόρεια Κύπρο ποια είναι η συσχέτιση αυτών των κυκλωμάτων με ε, την ε, εμπορία οργάνων, με όλες αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες. Τι να τους κάνουμε τους ωραίους νόμους αν κανείς δεν τους εφαρμόζει. Κυρία Σπινέλη. Να ευχαριστήσω τη συναδελφό Βαλερό για το, την εξαιρετική της δουλειά. Οι τροπολογίες που υπέβαλα θεωρώ ότι θα συμπληρώσουν το δικό της ε, σχέδιο γνωμοδότησης. Υπέβαλα τροπολογίες κατά κύριο λόγο που ζητώ την αναγνώριση ενός νέου είδους εμπορίας ανθρώπων για λόγους εκβιασμού που συχνά συνοδεύεται από βασανιστήρια στο ΣΥΝΑ και είναι αιτία πολλών δολοφολιών και εξαφάνισης ε, ερυθρέων προσφύγων ε, που έχουν απαχθεί. Όσοι επιβιώνουν από αυτή την τραυματική εμπειρία δεν λαμβάνουν συχνά την υποστήριξη στην Ευρώπη διότι η εμπορία αυτού του τύπου δεν αναγνωρίζεται επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την Ερυθρέα τον περασμένο Μάρτιο ανέφερε ήδη αυτού του είδους ε, το νέο τύπο εμπορίου και πρέπει, κατά να αναφέρουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση τη μορφή του και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται. Άλλες τροπολογίες της ομάδας μου υπενθυμίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς δασμολογικών προτιμήσεων επιπρόσθετων στις συμφωνίες με ορισμένες τρίτες χώρες για την προήθηση της επικύρωσης και της πραγματικής εφαρμογής των κύριων διεθνών συνθήκων για τα δικαιώματα, την εργασία, την προστασία του περιβάλλοντο. Επιπλέον, θα ήθελα, σας παρακαλώ, να γίνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλαμβάνει σε όλες τις ε, διεθνείς συμφωνίες της Ένωσης, ε, όπως και οι εμπορικές, οι επενδυτικές συμφωνίες που έχουν συναυθεί, που θα συναυθούν, δεσμευτικές ρήτρε αδιαπραγμάτευτες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εμπορία. Τέλος, υπέβαλα τροπολογίες για τη διάσταση του φύλου στο τομέα του εμπορίου, της εμπορίας ανθρώπου. Αναφέρω την αναγκαιότητα συνεργασίας, σοβαρής συνεργασίας δικαστικής μεταξύ των κρατών μελών και αναφέρω και την ανάγκη να αναγνωρίσουμε τις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν το θύμα της εμπορίας και το μετανάστη, τον πρόσφυγα ε, καταστάσεις που και στις δύο περιπτώσεις χρειάζονται υψηλά επίπεδα προστασίας και αποφυγή του επαναπατρισμού σε κράτη όπου υπάρχει κίνδυνος ε, οι πρόσφυγες να χάσουν τη ζωή τους ή να υποστούν φυσική, φυσικές επιπτώσεις, σωματικές επιπτώσεις. Ευχαριστούμε η εισηγήτρια κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω σε τρεις ερωτήσεις που ακούστηκαν η Τράπεζα Δεδομένων της Ευρωπόλ. Υπάρχει αυτή η πρόταση. Εμείς δεν συμφωνούμε όμως σε αυτό το σημείο μεταξύ μας, οπότε θα κάνουμε χωριστή ψηφοφορία. Διότι όπως φαίνεται δεν συγκλίνουν όλες οι απόψεις. Ε, ε, αλλά θα ψηφίσουμε έτσι, όπως είπαμε. Όσον αφορά την, το διαχωρισμό μεταξύ εμπορίας και διακίνησης, έχουμε ένα συμβιβασμό για αυτό το σημείο που αναφέρει ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση όπου κάποιος αφού διακινηθεί ε, στη συνέχεια γίνεται θύμα εμπορίας ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει ήδη επί ευρωπαϊκής επικράτειας και αυτή την περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη στις ε, συμβιβαστικές μας τροπολογίες και έτσι πιστεύω η διατύπωση που βρέθηκε να ικανοποιήσει άπαντες. Μετά το θέμα του ΣΥΝΑ. Πριν από ένα χρόνο περίπου συνάντησα για πρώτη φορά αυτό το ζήτημα και αποτελεί πρόβλημα. Το οποίο δεν έχουμε διαχειριστεί καθόλου στην πραγματικότητα. Η τροπολογία που έχουμε γι' αυτό ε, είναι νομικό ζήτημα ουσιαστικά έχει, να κάνει μάλλον περισσότερο με εξωτερικέ υποθέσεις παρά με εσωτερικέ. οπότε είναι δύσκολο να το συμπεριλάβω στη δική μου γνωμοδότηση για τη ΛΥΜΠΕ. Ωστόσο θα την ψηφίσουμε. κάποιε άλλε τροπολογίες που υποβλήθηκαν ε, αναγνωρίζεται περισσότερο ω τροπολογίε τη Επιτροπή Εξωτερικών ε, Υποθέσεων ε, ή αφορούν περισσότερο την ΤΡΟΑ και όχι εμά. Ωστόσο, μπορούμε να τι δούμε και να τι ψηφίσουμε, αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Βαλέρο. Η ψηφοφορία στη ΛΥΜΠΕ προβλέπεται για τις 28 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση αυτού του σημείου. Το επόμενο σημείο σήμερα το απόγευμα αφορά την οδηγία καταπολέμησης τη τρομοκρατία και αντικατάσταση τη απόφαση πλαισίου του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση τη τρομοκρατία αντικαθιστά η οδηγία του 2002 ε, παρουσιάστηκε στις 17 Μαρτίου και τώρα θα κάνουμε μια συζήτηση για τις τροπολογίες που υποβληθούν. Κυρία Χολμάιερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ πρώτα τους και όλους συζητητές οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε τρεις ε, μεγάλες συνεδριάσεις. Καταφέραμε σε αυτές τις τρεις συνεδριάσεις να έχουμε αρκετό χρόνο έτσι ώστε να συζητήσουμε με εμπειρογνώμονες οι οποίοι μας μετέφεραν την πραγματικότητα των κρατών μελών, μας μετέφεραν το τι συμβαίνει. Είχαμε καλέσει εισαγγελείς, δικαστές και ε, ενημερωθήκαμε. Είχαμε έναν Ιταλό εισαγγελέα την τελευταία φορά, ο οποίος ε, μας εξέθεσε με μεγάλες λεπτομέρειες το πώς ακριβώς η Ιταλία αντιμετωπίζει αυτά τα νέα δεδομένα της ε, καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας και αρκετές φορές ε, οφείλω να ομολογήσω ότι ε, μας πάγωσε το αίμα στις φλέβες με αυτά που ακούσαμε. Δεν πιστεύαμε ότι στον κόσμο υπάρχει τέτοια βαρβαρότητα, ιδιαίτερα με θύματα μικρά παιδιά από τους ε, τρομοκράτες. Πραγματικά μείναμε με κομμένη την ανάσα όση ώρα μιλούσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τους συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν πάνω από 400 ε, τροπολογίες. Ήταν εξαιρετική συνεργασία μας και οι τροπολογίες έχουν ως στόχο καταρχάς να, ε, να είναι συμβιβαστικές, να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος ε, θεμάτων, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο από το 2002 και το 2008, το οποίο έχει ε, στο μεταξύ ενσωματωθεί πλήρως στην νομοθεσία των κρατών μελών. Προσπαθούμε λοιπόν, ε, χρησιμοποιώντας αυτό, να ε, το συνδέσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε ορισμένες ε, παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, για παράδειγμα τα δεδομένα των επιβατών, τα PNR, συζητήθηκε το ε, θέμα των ε, υπηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγαίνουν στη Συρία ή στο Ιράκ και συμμετέχουν σε εκπαίδευση για τρομοκρατικές ε, δραστηριότητες. Το συζητήσαμε το τι θα κάνουμε όταν αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν πράξη αυτά για τα οποία εκπαιδεύτηκαν. Για παράδειγμα κάποιος από τη Γερμανία πάει στη Συρία, επιστρέφει, πετάει στη Ρώμη το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, δεν αφορά μόνο τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βρίσκεται μόνο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται εντός και η απειλή είναι μεγάλη. Σίγουρα πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε οι αποφάσεις οι οποίες περιέχονται στην Οδηγία για την Τρομοκρατία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προέρχονται από αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και του FATF. Έτσι, επομένως, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει χρησιμοποιήσει ε, την ε, διεθνή. Χθες, κατά τη συνομιλία με τον Ισαγγελέα, κατέστη σαφές ότι η υπάρχει ανάγκη για σωστή επικοινωνία, πρέπει να ε, τεθούν ε, σαφή όρια, πρέπει να προστατευτεί η ελευθερία των πολιτών και γι' αυτό χρειάζεται, ή μάλλον θα έλεγα πως είναι αναγκαία η ε, συλλογή αυτών αποδεικτικών των αποδεικτικων Προτού προβούν οι αρχές σε κάποια σύλληψη, έτσι ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να συλληφθεί κάποιος ε, άδικα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τα ε, σωστά αποδεικτικά στοιχεία, να υπάρχουν αποδείξεις προτού συλληφθεί κάποιος και οδηγηθεί στο δικαστήριο. Τώρα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελίε στα κράτη-μέλη έχει να κάνει με το εξή. Εάν θέλουμε να αποφύγουμε εγκληματικές ενέργειες μεγάλου βεληνικούς όπως τις Βρυξέλλες, όπως το Παρίσι, πρέπει να ε, φροντίσουμε, να συλλάβουμε τους ε, εγκληματίες προτού προβούν σε αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται μία ε, μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται να συλλεχθούν δεδομένα έτσι ώστε να μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτούς τους εγκληματίες πριν γίνει το κακό. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Στην Ιταλία πολλές φορές ε, συνάντησαν προβλήματα στη συλλογή αυτών των δεδομένων και η... αυτό που ακούσαμε χθες από τον εισαγγελέα με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να γίνει πραγματικότητα η σωστή συλλογή δεδομένων. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε και ε, να σταματήσουμε τους πιθανούς μελλοντικούς δράστες προτού δράσουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να αποτρέψουμε το έγκλημα πριν αυτό συμβεί, για να μην οδηγηθούμε πάλι σε εκατόμβες βεστημάτων. Αυτό όμως απαιτεί ε, την ε, σωστή συνεργασία και των πολιτικών και αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Ξέρετε, το χειρότερο είναι να έχει θύματα στην ίδια σου την οικογένεια από τέτοιες ε, ενέργειες. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαίρομαι πάρα πολύ που ήμασταν απόλυτα σύμφωνοι στο θέμα των ε, δικαιωμάτων των θυμάτων. Τα θύματα πρέπει και οι οικογένειες των θυμάτων δεν πρέπει να πληρώσουν δικαστικά έξοδα, πρέπει να τους παράσχεται νομική βοήθεια και κατά τη διάρκεια των ερευνών και στο δικαστήριο. Διαφορετικά τα θύματα δεν θα έχουν καμία βοήθεια. Επίσης πρέπει να ε, παρέχεται βοήθεια και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τώρα, η Ολλανδική Προεδρία είναι έτοιμη να αρχίσει τον τριμερή διάλογο από τον Ιούνιο και θέλουμε να προσπαθήσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το, το Κοινοβούλιο και ε, το Συμβούλιο να αρχίσουν ήδη από τον Ιούνιο έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ψηφοφορία τον Ιούλιο. Θέλουμε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο και ελπίζω το δυναμικό που έχουμε και η ορμή που έχουμε να συνεχίσει και στο τεμερή διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία το Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη συναδελφα Χολμάιερ για τις προσπάθειές της και για την επιλογή της μεθοδολογίας οι συναντήσεις των σκιωδών με εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες ε, και από διάφορους χώρους εργασίας ε, και που μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την αξιολόγηση και την εμβάθυνση είναι κάτι για μας πολύ σημαντικό. Διότι εμείς σήμερα έχουμε κληθεί να φέρουμε εις πέρα σε ένα κείμενο το οποίο σε όσους αντιμετωπίζουν καθημερινά επιτόπου αυτή τη δραματική μορφή εγκλήματος που είναι η τρομοκρατία. Καλούμαστε λοιπόν να τους παρέχουμε εργαλεία αποτελεσματικά. Με ικανοποίησε λοιπόν που το επενθύμισε και η Μόνικα αυτό ε, η συμβολή του εισαγγελέα Νικόλα Πιατσέντε. Ήταν μια σημαντική συμβολή και με ικανοποίησε αλλά γέννησε και ερωτηματικά ως προς το ποια θα ήταν τα καταλληλότερα μέτρα για να καλύψουμε τα κενά εκείνα που μερικές φορές ε, εμποδίζουν την αντιμετώπιση τόσο σημαντικών εγκλημάτων. Όπως γνωρίζουμε, το είπε και η συνάδελφος, έχουμε να κάνουμε μια τρομοκρατία διαφορετική από αυτήν που γνώριζαν οι χώρες μας μέχρι σήμερα, όπως και η δική μου η χώρα, η Ιταλία, αντιμετωπίζαμε μια τρομοκρατία εσωτερική, ενώ τώρα η τρομοκρατία προέρχεται από το εξωτερικό. Αλλά διαπράττει και από ανθρώπους με ευρωπαϊκά διαβατήρια που ζουν στις χώρες μας. Και έχει μορφές νέες και ιδιαίτερα περίπλοκες. Καθήκον μας λοιπόν ε, είναι κάτι πολύ ευαίσθητο και έχουμε μια τεράστια ευθύνη διότι καλούμαστε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της διαφύλαξης των κεκτημένων δικαιωμάτων όπως η ελευθερία κίνησης, μετακίνησης και των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας ε, για τους πολίτες το δικαίωμα για την ελευθερία και το δικαίωμα για τη ζωή ε, πρέπει ε, να τα χειριζόμαστε με τον ίδιο σεβασμό. Οπότε θα πρέπει στο κείμενό μας ε, να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των απαιτήσεων. Μα υπενθυμίζετε εδώ ότι όταν έγινε η απόφαση πλαίσιο κατά τη τρομοκρατία, το Κοινοβούλιο δεν είχε τι σημερινέ αρμοδιότητε ε, όπω το αναγνωρίστηκαν από τι συνθήκε Λισαβόνα. Γι' αυτό το λόγο, εγώ πιστεύω ότι σήμερα έχουμε μια μεγαλύτερη σημαντική ευθύνη ενώπιον ενός, ε, μια τρομοκρατία που ξαφνικά εκδηλώνεται όπω είδαμε και όπω είπαμε, όπω είδαμε και δίπλα μα ε, στην πόλη μα, δίπλα στο κοινοβουλίο μα, με μορφέ, πραγματικά δραματικέ. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται πραγματικά να δουλέψουμε εξετάζοντας προσεκτικά τις διάφορες πτυχές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εγκλημάτων που εμείς θέλουμε να εντοπίσουμε. Οι τροπολογία των διαφορών ομάδων, ε, υπέβαλε και η δική μου ομάδα φυσικά, προφανώς ε, ε, καταδεικνύουν θέσεις πολύ απομακρυσμένες μέχρι στιγμής. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όπου είναι δυνατόν και συμμερίζομαι την επιλογή της εισηγητρίας, όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες και μετά να εμβαθύνουμε τα θέματα αυτά που σήμερα μας διαχωρίζουν, αλλά που είναι θέματα βέβαια εξαιρετικά περίπλοκα. Ε, η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων ε, δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο, ειδικότερα το πρωτόκολλο το, προς το πρωτόκολλο της συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η ελάχιστη επέτηση. Δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε, αλλά κάθε επιλογή θα πρέπει να ζυγιστεί σωστά. Και να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα το θέμα των ταξιδιών για τρομοκρατικούς σκοπούς. Ένα θέμα που έχει πολλές πτυχές. Υπάρχουν διεθνείς νομοθεσίες ε, για τη ροή των μαχητών στη Συρία και στο Ιράκ, αλλά σήμερα έχουμε διαφορετικά φαινόμενα. Έχουμε τους ε, επαναπατρισμένους ε, μαχητές ε, δικούς μας υπηκόους και όσους έρχονται στην Ευρώπη για να διαπράξουν τρομοκρατικές ε, ενέργειες ή για να δικαστούν σε μια χώρα και όχι σε άλλη. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και τους διάφορους τύπους τους. Αλλά υπάρχει και άλλη μια πτυχή ε, για την οποία συμμερίζομαι τόσα είπε συνάδελφος. Η αυτό που έχει προσδιοριστεί και το βλέπουμε όλοι, αυτό που έχει προσδιοριστεί από τον εισαγγελέα τον κ. Πιατσέντη. Τα γεγονότα στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες ε, αποτελούν μάλιστα την απόδειξη, διότι διαπράχθηκαν από ε, ανθρώπους που είχαν ποινικό μητρό. Όπως υπενθύμισε λοιπόν ο συνάδελφος, ο Δ. Πιατσέντινη μας ε, είπε ότι στην Ιταλία έχουν καταλήξει στο να κλείνουν έρευνες πολύ σημαντικέ για το οργανωμένο έγκλημα ή για την τρομοκρατία ε, και έφεραν καλά αποτελέσματα διότι λειτουργήσαν καλά υπηρεσίε πληροφοριών συλλέγοντας πληροφορίες ε, πριν την έρευνα αλλά που έπαιξαν θεμελιωδή ρόλο για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα. Πέραν λοιπόν των δικών μας εργασιών ε, σύνταξη των διαφορών άρθρων που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε με την αναφορά του στα ταξίδια, στην πρόσληψη, στις, στη στρατολόγηση μέσω διαδικτύου. Μας το είπε και ο κύριος Πιατσέντη, να δούμε τις μορφές ε, αυτοεκπαίδευσης, αυτοστρατολόγησης και όλα αυτά αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις να έχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών, αστυνομικών υπηρεσιών και δικαστικών υπηρεσιών, διότι η έγκυρη ανταλλαγή πληροφοριών, επαρκών πληροφοριών, αποτελεί βασική προϋπόθεση, χωρίς την οποία όσο καλή και να είναι η νομοθεσία που ελπίζω εμείς να καταφέρουμε να συντάξουμε, δεν θα μπορέσει να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε από πλευρά μου θα συνεχίσουν να είμαι διαθέσιμη για συνεργασία ώστε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια καλή ισορροπία μεταξύ των διαφορών απαιτήσεων και των διαφορών δικαιωμάτων και να γράψουμε ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης των δραματικών μορφών τρομοκρατίας που παρατηρούμε τελευταία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντεπρέ που αντικαθιστά τη και Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τον κύριο Τσέζεκ αντικαθιστώ εγώ, ο οποίος ε, ζητώ συγγνώμη που είχε ανελημμένες υποχρεώσεις. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα σας διαβάσω το κείμενο του κύριου Τσέζεκ, με το οποίο συμφωνώ και εγώ προσωπικά. Παρόλο που γνωρίζω ότι κάποιοι προσανατολισμοί σήμερα συζητιούνται έντονα και μέσα στην δικιά μου την ομάδα. Εγώ συμφωνώ πάντως μαζί με τον κύριο Τσέζεκ, γι' αυτό και θα σας ε, διαβάσω τις παρατηρήσεις τους έχουν. Στόχος του κειμένου είναι να πετύχουμε σε μια κοινή βάση ποινικών κυρώσεων όταν πρόκειται για εγκληματικές πράξεις ή όταν πρόκειται για ένα πρώτο βήμα για την δίωξη μιας εγκληματικής ε, πράξης. Ο κύριος Σεζέκ συνεχίζει λέγοντας «Πρέπει να συμφωνήσουμε καταρχήν για αυτό το οποίο αποτελεί μια προπαρασκευαστική πράξη για να συμμετάσχει κανείς σε μια τρομοκρατική ενέργεια που αναφέρονται ως παραβιάσεις σχετικές με τρομοκρατικές πράξεις στο κείμενο. Ο κύριος Σεζέκ πιστεύει επίσης ότι δεν δίνουμε όλη την ίδια σημασία σε αυτές τις πράξεις. Γι' αυτό και για μένα είναι σαφές ότι η δημοσίευση ε, μηνυμάτων τα οποία οθούν στο μίσος ή άλλες μέθοδοι που οθούν σε τρομοκρατικές πράξεις ή στο να συμμετάσχει κανείς σε μια τρομοκρατική ομάδα ή να προβεί σε μια τρομοκρατική πράξη, όλα αυτά αποτελούν προπαρασκευαστικές δράσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη. Λέει, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες θέλουν να διαγραφούν κάποιες από τις δράσεις αυτές που απαριθμούνται προς ποινική δίωξη. Δεύτερον, το άρθρο 15 είναι ένα άλλο βασικό σημείο για τον κύριο Σέζεκ αλλά και για μένα. Για να μπορέσουμε να διώξουμε έναν ε, υπεύθυνο, δεν πρέπει να περιμένουμε να λάβει χώρα η τρομοκρατική ενέργεια. Είναι βασικό, αν θέλουμε να επιτρέψουμε στις κατασταλτικές αρχές, να είναι αποτελεσματικές. Άπαξ και ένα άτομο πηγαίνει να καταρτιστεί, να συμμετέχει σε μια τρομοκρατική ομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι συγκεκριμένο το σχέδιό του για μια τρομοκρατική επίθεση. Θα πάρει όμως πληροφορίες κάποια στιγμή και το να επιβάλλουμε στις αρχές να αποδείξουν ότι το συγκεκριμένο άτομο σκοπεύει να προβεί σε συγκεκριμένη ε, τρομοκρατική επίθεση δεν είναι κάτι κατάλληλο για αυτό το κείμενο. Τέλο ο κ. Σίκε λέει δεν μπορώ να στηρίξω τι τροπολογίε που βγαίνουν προ αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Σχέτε, θέλω να επιμείνω τώρα και να σχολιάσω κάποιε τροπολογίε που έχουν υποβληθεί και που όλε έχουν σαν στόχο τη βελτίωση τη ε, πληροφορία και το πώ οι πληροφορίε αυτέ θα αντιμετωπίζονται πιο συστηματικά. Πιστεύουμε ότι οι χώρε μέλη πρέπει συστηματικά να συμπεριλαμβάνουν στο ΣΥΣ κάθε άτομο το οποίο υποπτεύονται που έχει προχωρήσει σε παραβιάσεις βάση του 3414 και τις περοπαρασκευαστικές ανέργειες. Οι χώρες μέλη έχουν την υποχρέωση επίσης να ενημερώνουν την Europol για κάθε ύποπτο όσον αφορά τις παραβιάσεις που αναφέρονται στα σημεία 314. Επίσης, κυρία Πρόεδρε και κυρία Συγγήτρια, Θέλουμε οι χώρες μέλη και είχαμε την ευκαιρία όλοι να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να ανταλλάσσουν όλα τα στοιχεία PNR σε σχέση με ύποπτους ή άτομα που έχουν καταδικαστεί για μία από τις παραβιάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3-14 της παρούσης οδηγίας. Εγκρίναμε την PNR βάσει ε, του κειμένου αυτού τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση. Είναι όμως οτική σημασία. Η οδηγία έχει ως συγκεκριμένο στόχο την εναρμόνιση των πρακτικών για να καταπολεμηθούν οι προπαρασκευαστικές δράσεις και οι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι συνεπώς αναγκαίο οι χώρες μέλη να ενημερώνουν, να κοινωνούν δηλαδή στις άλλες αρχές τα στοιχεία PNR που έχουν να κάνουν είτε με υπόπτους είτε με άτομα που έχουν καταδικαστεί σε σχέση με την τρομοκρατία. Και κάτι ακόμα και θα τελειώσω με μια ερώτηση. Ο τίτλος που δώσαμε προβληματίζει την ε, Επιτροπή, αλλά μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τελειώνω με το εξή. Κάθε κράτο μέλο πρέπει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αντιμετωπίζει τις παραβιάσεις που αναφέρονται σε άρθρο 314 εφόσον ο, το άτομο βρίσκεται στην επικράτειά σας. Μπορείτε στη χώρα σας να διώξετε κάποιον που είναι της δικιάς σας υπηκότητας είτε κάποιον άλλης υπηκότητας που όμως ε, προχωράει σε δράση η οποία τιμωρείται ποινικά στη χώρα σας. Τώρα, αν στην επικράτειά σας είναι κάποιο που έρχεται από τρίτη χώρα, ο οποίο έχει προβεί σε παραβίαση στη χώρα σας και μπορεί να μην είναι γνωστό αμέσως, αλλά να το μαθαίνετε κατά τη διάρκεια κάποιας άλλης έρευνας. Θέλουμε στην περίπτωση αυτή να συζητήσουμε τη δυνατότητα, την αρμοδιότητα δίωξης του ατόμου αυτού να τη δώσουμε στο κράτος αυτό στο οποίο έγινε η πράξη, ακόμα κι αν το άτομο αυτό δεν έχει την επικότητα της χώρας όπου έγινε η τρομοκρατική αυτή πράξη, ακόμα και αν η τρομοκρατική αυτή πράξη έχει λάβει η χώρα κάπου αλλού, αλλά το άτομο βρίσκεται στην επικράτειά σας. Κυρία Φεράρα, ευχαριστώ πολύ να μιλήσω εκ μέρους της συναδέλφου Λαρατζέα που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για λόγω άλλων δεσμεύσεων, οπότε θα σας διαβάσω τα όσα θέλει να σας διαβιβάσει να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις εργασίες της και τη δέσμευση των συναδέλφων με τις που με τις τροπολογίες βελτιώνουν την πρόταση. Ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών αναδεικνύει την το πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Υποστηρίζω τις τροπολογίες ε, που αφορούν τα χαρακτηριστικά των ε, εγκλημάτων και σίγουρα με την ποινικοποίηση ορισμένων συμπεριφορών όπως το ταξίδι και την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών λέω ότι θα πρέπει να βασίζονται σε νομικές αρχές και βάσει στοιχείων αντικειμενικά επαληθεύσιμων ε, δεν μας ικανοποιούν οι περιορισμοί των ε, ελευθεριών ε, στο, έκφραση στο δίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε δεν θα υποστηρίξουμε αυτές τις τροπολογίες. Ξέρετε, το δίκτυο μπορεί να μετατραπεί σε μέσο ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τρομοκρατών και να διευκολύνει τη ριζοσπαστικοποίηση. Γι' αυτό το λόγο ζητάμε Κάθε παρέμβαση περιορισμού στο διαδικτύο να συνοδεύεται από κάποιον αυτόνομο έλεγχο της δικαστικής αρχής. Θα αναλάβουμε την ευθύνη ώστε πτυχές σημαντικές όπως η πρόληψη των τρομοκρατικών ενεργειών και της ριζοσπαστικοποίησης να αναδεικνύονται σωστά στην οδηγία. Η πρόληψη πρέπει να συνοδεύεται από κατασταλτικές ενέργειες αναγκαστικά διαφορετικά. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα θεωρηθεί χαμένη υπόθεση από την αρχή. Κάτι άλλο σημαντικό είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανάγκη ενίσχυσης και της αστυνομική συνεργασίας υποχρεωτικά και της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Όπως και άλλες, ε, άλλοι συνάδελφοι άλλων ομάδων θεωρούμε ότι η οδηγία με την οποία ασχολούμαστε σήμερα πρέπει να περιλαμβάνει ε, αναφορά σε αυτή τη συνεργασία και στον υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Θέλουμε επίσης να συμπεριλάβουμε μια αναφορά στο διαχωρισμό των τρομοκρατικών ομάδων. Από την Ιταλική εμπειρία μπορούμε να προσδιορίσουμε τα μοντέλα. Ε, στη χώρα μου έχουμε καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και έχουμε εμπειρία σε αυτό, οπότε θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν συστήματα και προγράμματα προστασίας όσων συνεργάζονται με τις αρχές για την ευκολότερη αποσάρθρωση των τρομοκρατικών δικτύων και για να ε, βρίσκει δικαιοσύνη τους εγκληματίες ε, και να προλαμβάνονται νέες τρομοκρατικές ενέργειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φεράρα. Κυρία Σπινέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να επιστήσω ξανά την προσοχή της εισηγήτριας στην γερμανική νομολογία, η οποία μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα όσον αφορά την νομοθεσία καταπολέμησης της τρομοκρατίας μέσω του Bundeskriminalamt και του Γραφείου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Ε, φανταζόμαι ότι η συνάδελφος κ. Χόλμα γνωρίζει άριστα αυτή την ομολογία και έχω στο νου μου την απόφαση της 20 Απριλίου, δηλαδή χθες του δικαστηρίου, όπου επιβεβαιώνεται ότι η νομοθεσία σε μεγάλο βαθμό είναι αντισυνταγματική. Ειδικότερα είναι αντισυνταγματική η παρακολούθηση και οι τηλεφωνικές υποκλοπές και τα μέτρα τα οποία δυσανάλογα εφαρμόζονται ε, στην ιδιωτική ζωή των ε, πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι ε, τα εθνικά δικαστήρια μας ε, κάνουν κάποια πολύ καλά μαθήματα σε εμάς τους Ευρωπαίους νομοθέτες. Μαθήματα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας, να υπενθυμίσω ότι ήδη δύο φορές ε, τα γερμανικά δικαστήρια αμφισβήτησαν ε, νόμους που έχουμε συζητήσει ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω στο νόμο τώρα το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης και την Προστασία Δεδομένων. Γιατί είναι καλό αυτό το μάθημα, διότι αν η δική μας οδηγία είναι υπερβολικά ασαφής όσον αφορά το κράτος δικαίου και ε, επεμβαίνει υπερβολικά στην ιδιωτική ζωή, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ένα εθνικό ή ευρωπαϊκό δικαστήριο να αναφέρει σε κάποια στιγμή την αρχή της αναλογικότητας των νόμων μας. Ευχαριστώ. Thank η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πρέπει να βρούμε σε μια σύγκληση σε αυτήν την οδηγία και πιστεύω πως μπορούμε να τα βρούμε. Χαίρομαι που βλέπω ότι καταβάλουμε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτή την οδηγία για μένα είναι σημαντικό να δείξουμε ότι Είμαστε διαφορετικοί από τους τομοκράτες. Σεβόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ορίσουμε με σαφήνεια τον ε, σκοπό, την πρόθεση τέλεσης εγκληματικής ενέργειας. Και θα ήθελα να πω ότι το κλειδί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις τράπεζες δεδομένων, το, τη δικαστική εξουσία, τις αστυνομικές αρχές και την ανταλλαγή απόψεων ε, μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Αλλά και διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις ε, πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα δίκτυα πληροφοριών και στις αστυνομικές αρχές. πολλές φορές συχνά είναι στο εθνικό επίπεδο το πρόβλημα, όχι στο ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό χρειάζεται να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να μαζέψει τα κράτη-μέλη, να τα καλέσει στην τάξη. Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα χάλι. Πρέπει να προσέξουμε τα όσα μας είπαν οι εμπειρογνώμονες. Υπάρχει ξεκάθαρη διασύνδεση ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα ε, και ε, σε όσους στρατολογούνται, μικροεγκληματίες στρατολογούνται για να διαπράξουν τρομοκρατικές ενέργειες. Είδαμε και στην έκθεση Ντάτη εξάλλου πώς οι φυλακές, αντί να είναι σοφρονιστικά ιδρύματα, είναι κέντρα ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε ότι αυτοί που μας επιτέθηκαν δεν είναι ξένοι μαχητές. Είναι δικοί μας εδώ ντόπιοι μαχητές και μάλιστα τα περισσότερα θύματα ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν μουσουλμάνοι. Τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε κατάσταση άρνησης, αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι το πρόβλημα βρίσκεται εντός και όχι εκτός. Και πολύ συχνά οι θήτες έχουν υπάρξει θύματα κακής πολιτικής ένταξης, κακής οικονομικής πολιτικής ε, περιθωριοποίησης που έχει οδηγήσει σε πάντως είδους ε, εκτροχιασμούς με τα γνωστά αποτελέσματα, τη στρατολόγηση. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω με αυτήν την οδηγία να διορθώσουμε ένα μεγάλο λάθος, το PNR. Σε αυτό αναφέρομαι. Δεν πιστεύω πως αυτό ήταν η ασημένια σφαίρα που θα έλυνε όλα τα προβλήματα. Σίγουρα είναι ένα εργαλείο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί και να αποβεί χρήσιμο, όμως τώρα κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Και αυτό διότι οι κυβερνήσεις μας δεν ήθελαν ένα ενοποιημένο σύστημα για τις πτήσεις τσάρτερ για τις ιδιωτικές πτήσεις, οι οποίες μάλιστα απουσιάζουν από το σύστημα PNR. Και η χρηματοδότηση, ξέρετε, της τρομοκρατίας πολύ συχνά συνδέεται με ε, εγκληματικές δραστηριότητες παντός τύπου. Διότι χρειάζονται πόρους ε, ιδιωτικά αεροσκάφη, τα πάντα. Χρησιμοποιούν τα πάντα για να πετύχουν το σκοπό τους και γι' αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο, είναι εξοργιστικό ότι υπάρχουν τέτοια παραθυράκια στο PNR. Η κυρία Εντφέλντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Ε, πρώτα απ' όλα έχω αμφιβολίες για το όλο σκεπτικό της ποινικοποίηση ε, ταξιδιού με ε, σκοπό την τρομοκρατία. Η ποινικοποίηση των προθέσεων είναι κάτι το πάρα πολύ επικίνδυνο. Άλλο η ποινικοποίηση της πράξης και άλλο της πρόθεσης. Και η κυρία Χολμάιερ πολύ σωστά είπε ότι χρειάζονται αποδείξεις. Πώς λοιπόν θα αποδείξεις τις προθέσεις κάποιου. Και εδώ έρχομαι στο ουσιαστικό κομμάτι, στο, στο πρακτικό θέμα. Πολλοί νέοι ταξιδεύουν σε μέρη όπως Συρία, Ιράκ κτλ αυτοί οι νέοι είναι επιρρεπείς σε μηνύματα πάντως τύπου. Και μετά όταν φτάνουν εκεί συνειδητοποιούν ότι έχουν κάνει λάθος. Και όταν το συνειδητοποιούν επιστρέφουν. Εάν λοιπόν τους ποινικοποιήσουμε, τι θα συμβεί. Δεν θα τους βοηθήσουμε να ε, ξεφύγουν. Όπως είπε και η κυρία Γκόμες, αν τους ε, βάλει στη φυλακή, ο κίνδυνος να βγουν από τη φυλακή ε, τρομοκράτες είναι μεγαλύτερος από το να σοφρονιστούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που συμμετέχουν σε προγράμματα από με μεγάλη επιτυχία και πιστεύω πως αν χάσουμε την ε, ευκαιρία θα κάνουμε μεγάλο λάθος. Γι' αυτό λοιπόν οι λόγοι δεν είναι μόνο αρχής αλλά είναι και πρακτικοί. Έπειτα, κάτι που είχα αναφέρει και στην αρχική συζήτηση για την πρόταση, είναι ότι εμείς εδώ δεν νομοθετούμε βραχυπρόθεσμα. Θέλουμε να νομοθετήσουμε μακροπρόθεσμα και στοχεύουμε συγκεκριμένα είδη τρομοκρατίας. υπάρχουν ακροδεξιές ομάδες στις χώρες μας οι οποίες μπορούν να πηγαίνουν από τη μία πόλη στην άλλη με λεωφορείο, με σκοπό τρομοκρατικές ενέργειες. Αλλά εμείς από ό,τι, παρατηρώ εφαρμόζουμε ε, τον ορισμό της τρομοκρατίας μόνο σε ορισμένες ομάδες. Δεν είναι μόνο οι Ισλαμιστές, ξέρετε, που διαπράττουν τρομοκρατικές ενέργειες για να διαταράξουν τη δημοκρατία για μένα έχουν... Για μένα αυτοί είναι ε, τρομοκράτες, αλλά τρομοκράτες είναι και άλλοι που δρούν εντός της χώρας τους. Γι' αυτό λοιπόν, εάν νομοθετήσουμε χωρίς... Ε, εάν νομοθετήσουμε στοχεύοντας μια συγκεκριμένη ομάδα, ε, θα αφήσουμε μια άλλη ελεύθερη. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί ε, σχετικά με το πώς νομοθετούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι Ισπανίδα, λέει η κυρία Μπαγκαρφατουάτ Ρουίτ. Ξέρουμε τι σημαίνει ριζοσπαστικοποίηση, βία, επιθέσεις. Έχουμε περάσει πολλές και από περιφερειακές ε, τρομοκρατικές οργανώσεις και από τη διεθνή τρομοκρατία. Τώρα, όσον αφορά τα ταξίδια, διάβασα τις τροπολογίες και θέλω να σας πω το εξή. Ε, φυσικά, οι δοκιμές ε, που κάνουν οι τρομοκράτες φυσικά και πρέπει να ληφθεί υπόψη και οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκονται υπό, δικαστική, υπό δικαστικό έλεγχο. Αλλά όσον αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία, όταν μιλάμε για τα ταξίδια, να λάβουμε υπόψη μας ότι το ταξίδι γίνεται και εμείς από αυτό θα συμπεράνουμε ότι ανήκει σε μια τρομοκρατική οργάνωση ή ε, είναι, ανήκει σε μια τρομοκρατική ομάδα. Κάποιος ο οποίος έχει ριζοσπαστικοποιηθεί ή ήμι ριζοσπαστικοποιηθεί και αποφασίζει να πάει από μόνος του είναι κάτι διαφορετικό. Αν το ταξίδι γίνεται γιατί ανήκει σε μια τρομοκρατική οργάνωση, υπάρχει ήδη συνεργασία, είναι κάτι διαφορετικό. Το ότι ανήκει ή συνεργάζεται το άτομο μπορεί να μας χρησιμεύσει περισσότερο για να καταλάβουμε τι σημαίνει το ταξίδι. Γιατί μπορεί να πρόκειται για freelance. Τώρα, για την ποινική δίωξη υπάρχει το θέμα της συμμετοχής ή της συνεργασίας σε τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι το ίδιο σοβαρό όπως η συνεργασία σε μια δολοφονία ή δολοφονία. Υπάρχουν διαβαθμίσεις αλλά σε πιο χαμηλό επίπεδο ζημιάς προς την κοινωνία είναι η, πώς το, πω, το να είναι κανείς κοντά στην τρομοκρατία. Και αυτό ποινικοποιείται. Λοιπόν, για τα ταξίδια να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ποια γεγονότα έχουν λάβει χώρα και έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώνουν τις ελευθερίες μας η δικαστική, ο δικαστικός έλεγχος έτσι καλλιώς πρέπει να υπάρχει πάντα κάθε φορά που υπάρχει αστυνομική έρευνα. Αυτό έχω να πω σε Ισπανίδα. Ευχαριστούμε. Κύριος Φως. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που έχουμε ενώπιόν μας είναι οι συνέπειες των επιθέσεων είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να θεωρούμε μεμονωμένο περιστατικό, πρέπει να θεωρούμε μόνιμο συνοδό της ζωής μας. Αυτή είναι μόνιμη απειλή. Αυτήν την μάχη κατά της τρομοκρατίας, κατά του θρησκευτικού φανατισμού, όπως θέλετε πείτε το, δεν θα την κερδίσουμε εάν με μισή καρδιά προσπαθούμε εδώ να νομοθετήσουμε. Δεν πρέπει ε, να γίνει αυτό, διότι έτσι υπονομεύεται η ελευθερία που απολαμβάνουμε στην κοινωνία μας, έτσι υπονομεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, διότι ε, εάν επενδύσουμε σε τεχνογνωσία, σε προσωπικό, σε ε, τεχνολογία, τότε θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Καταρχάς, προληπτικά, ε, να προλάβουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έπειτα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για ε, όσους ε, ασχολούνται με τις, ε, για, τις αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν να προλάβουν κάποια ε, τρομοκρατική επίθεση. Αυτό χρειάζεται συλλογή πληροφοριών για να προλάβουμε να απομακρύνουμε τους τρομοκράτες πριν χτυπήσουν. Εδώ ποιο είναι το δύσκολο. Το δύσκολο είναι να φιλτράρουμε τα χρήσιμα από τα μη χρήσιμα. Να προστατεύσουμε τα δεδομένα που πρέπει να προστατεύσουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται και η δυνατότητα εδώ να ε, μπορούμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό, υπάρχουν πολλά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ε, αποκτήσουμε τις πληροφορίες και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης, είδαμε και στο, στη Συμφωνία SWIFT και στην FTP και στα PNR ότι θέλαμε να συνεργαστούμε με ε, διάφορα άλλα συστήματα έτσι ώστε να συνθέσουμε τα δεδομένα και να ε, οδηγηθούμε στο σωστό ε, αποτέλεσμα, στη σωστή πληροφορία. Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στις τράπεζες πληροφοριών πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο οριζόντιος τρόπος ε, που ε, διεξαγόταν η ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι τώρα ε, δεν έχει λειτουργήσει όπως θα έπρεπε διότι μας λείπουν οι γνώσεις. Όπως είπε και η Άννα Γκόμες, χρειάζεται να δώσουμε βάση στη διαλειτουργικότητα αυτών των βάσεων δεδομένων. Γι' αυτό χρειάζεται μία κεντρική υπηρεσία που να έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις ε, βάσεις δεδομένων, σε όλες τις πληροφορίες. Τώρα δεν είναι, ε, πιστεύω, σημαντικό να αποφασίσουμε Πώ θα οργανωθεί αυτό, ποιο θα είναι ο υπεύθυνο αν θα είναι ένα κρατό μέλο οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές κτλ. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν αυτές οι διασυνδέσεις και να υπάρχει και αυτή η κεντρική ε, πρόσβαση. Γι' αυτό χρειάζεται μια οδηγία που να αναφέρεται σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας, όπως αναφέρθηκε. Πρέπει να είμαστε στη θέση να ε, ανακαλύψουμε ποιος ε, ε, θέλει να κάνει μια τρομοκρατική ενέργεια, γιατί, πώς και χρειάζονται τα αποδεκτικά στοιχεία, τα οποία φυσικά θα συλλέξουμε στα πλαίσια του κράτους δικαίου, έτσι ώστε να μπορούμε να απομακρύνουμε αυτόν τον υποψήφιο τρομοκράτη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την σωστή συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, γι' αυτό και χρειάζεται πέραν ε, των υπολείπων που σας είπα και η σωστή κατάρτιση του προσωπικού, διότι ε, η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα όχι μόνο για μας αλλά και για τους τρομοκράτες. Ξέρετε, είναι πολύ... Ε, ε, είναι διασυνδεδεμένοι μέσω του διαδικτύου. Χρησιμοποιούν και αυτή τις τελευταίες τεχνολογίες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αυστηροί, ταχύτατοι και ε, να έχουμε συνοχή, διότι μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο και όχι να τον χάσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φώση. Κυρία Ζήπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, αλλά θα συνεχίσω στα γερμανικά. Με εκπλήσει η ελαφρότητα με την οποία αναφέρεστε εδώ στην ε, τράπεζα δεδομένων, στη βάση δεδομένων, ότι οι διασυνδέσεις πρέπει να είναι οριζόντιες, κάθετες, διαγώνιες. Με εκπλήσει αυτό. Καταρχάς υπάρχουν και νομικά όρια. Υπάρχουν νομικά όρια τα οποία μπορείτε να τα δείτε αν ε, κοιτάξετε τον τρόπο με τον οποίο στις νομικές αρχές επεξεργάζονται τα αιτήματα ασύλου. Έπειτα υπάρχει θέμα αρμοδιότητας. Δεν μπορεί ο καθένας να διαχειρίζεται δεδομένα και να έχει πρόσβαση σε αυτά. Τρίτον, η υποψία ε, κάποιου για την ριζοσπαστικοποίηση δεν φτάνει. Εντάξει, όταν, όταν υπάρχει υποψία ότι κάποιο έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, πρέπει φυσικά να αντιδράσει, όμως στα πλαίσια του νόμου. Οι αστυνομικές αρχές πρέπει να ε, δράσουν για την πρόληψη της ρίζοσπαστικοποίηση, αλλά υπάρχουν όρια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως πρέπει οι αρχές να είναι καταρτισμένες. Κύριος Μπόνι έχει το λόγο. Θα μιλήσω πολωνικά. Ε, λοιπόν, η τρομοκρατική απειλή θα συνεχίσει να αυξάνεται και το πρόβλημα συνιστάται στο εξή ερώτημα. Η οδηγία αυτή θα μα ε, βοηθήσει να, στην πρόληψη αυτών των δράσεων, γιατί η πρόληψη είναι το κλειδί. Δεν μπορούμε απλά να αντιδράμε σε πράγματα που έχουν ήδη συμβεί. Για να έχουμε σωστή πρόληψη χρειαζόμαστε έναν ευρύτερο ορισμό των εγκληματικών πράξεων, εγκληματικών πράξεων που οδηγούν σε ε, εγκληματικέ ενέργειες ε, στη χώρα μου, στην Πολωνία. Πολλοί αμφιβάλλουν κατά πόσο η οδηγία θα επιλύσει προβλήματα, οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε και γιατί έχει συνταχθεί με αυτόν τον τρόπο αυτή η οδηγία. Διότι θα καταστήσει δυνατό για τις αστυνομικέ αρχές να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση πολέμηση τη τρομοκρατία των τρομοκρατών και των πιθανών τρομοκρατών. Μετά τίθεται το ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι πολύ κρίμα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει τέτοια βούληση για ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, αν την καταστήσουμε υποχρεωτική, τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι ε, συμφωνήσαμε τη δέσμη μέτρων για την προστασία δεδομένων και αυτή η οδηγία, μια από αυτές τις οδηγίες, λέει σαφώς ποια είναι η βάση ε, πρόσβαση σε ορισμένου τύπου δεδομένων από την αστυνομία. Οπότε, ναι, μα ενδιαφέρουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ζητήσουμε και κάποια υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Βίδεμπερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αναφερόμαστε εδώ στο ε, δικαιώματα και στις ελευθερίες. Ε, εγώ δεν βλέπω αυτό το δικαίωμα ελευθερίας τι γίνεται τελικά ε, και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε 5.000 αλλοδαπούς μαχητές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλοδαποί μαχητές foreign fighters οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Έχουν ευρωπαϊκή υπηκότητα. Ε, πάνε και κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες ε, ή ε, κάνουν εγκληματικές ενέργειες, πρέπει να τους αφαιρούμε την υπηκότητα. Αυτό σημαίνει ασφάλεια, να προστατευτούμε, να μπορούμε να προστατευτούμε από ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν από τη Συρία. Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια, πρέπει να έχουμε σύνορα και ελέγχους. Δεν μπορούν αυτοί να μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Έτσι. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη προστασία. Δεν αρκεί το να άρα θέλουμε και μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά τι έρευνες, την ανταλλαγή πληροφοριών γνωρίζουμε ότι ήδη έχουμε πολλά η κόσμο που έχει επιστρέψει από τη Συρία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η Μόνικα. Σας ευχαριστώ πολύ ε, όλες και όλους σας για τη συνεισφορά και για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείξατε. Πιστεύω πως ε, οι παρεμβάσεις σας και μόνο δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον σας και πόσο σας ε, ενδιαφέρει να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Θα απαντήσω τώρα σε καθένα από σας, ε, αγαπητή κύριε Ντφέλντ. Αυτός ο νέος που συνελήφθη, συνελήφθη γιατί. Για τον σκοπό για την ιδιότητά του ταξιδιώτη, για το γεγονός ότι ταξίδεψε σε μέρος που ήταν ύποπτο και για το παρελθόν του ως Αυτό τον ε, καθιστά ύποπτο για πιθανές ε, για προθέσεις τρομοκρατικής ενέργειας. Γι' αυτό συνελήφθη. Και όταν τον συνέλαβαν δεν ήξεραν εάν όντως είναι ένας από αυτούς τους ε, ιδιαίτερα επικίνδυνους τρομοκράτες ή όχι, αλλά τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι υπήρχαν ε, βίντεο, υπήρχαν ε, αποδεικτικά ε, στοιχεία ότι προσπαθούσε να ριζοσπαστικοποιήσει τα παιδιά του. Τα παιδιά των ήταν 2 και 4 ετών. Ξέρετε τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Πώς ριζοσπαστικοποιούνται μικρά παιδιά, μωρά. Αυτό Λοιπόν, δεν φαινόταν από την αρχή. Δεν μπορούσαν από την αρχή να τον ε, καταδικάσουν για κάτι τέτοιο. Εάν όμως δεν τον είχαν συλλάβει, δεν θα είχαν το χρόνο να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία και να τον καταδικάσουν και να τον βρουν στο κάτω-κάτω. Αυτό έσωσε ζωές, ξέρετε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, αλλαγής. Και όπως είπε και ο Άξελ ή η Κατερίνα, Φυσικά και κανείς δεν θέλει να συλλαμβάνονται άνθρωποι και να ε, μπαίνουν στη φυλακή έτσι αυθαίρετα. Όχι, πρέπει πρώτα να συλλέγονται αποδείξεις. Εάν οι αποδείξεις μας δείξουν ότι πρέπει πρώτον ε, να παρουσιαστεί ο ύποπτος ενώπιον δικαστηρίου και δεύτερον εάν οι αποδείξεις μας δείξουν ότι όντως έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα και ε, να δούμε τη φύση του και να καταδικαστεί τότε μπορούμε να προλάβουμε ε, το, τα χειρότερα. Μπορούμε να προλάβουμε κάτι στην αρχή του και αντί για την φυλακή να ε, στείλουμε αυτόν τον άνθρωπο σε κάποιο... Ε, σε κάποια εναλλακτική ισοφρονιστική λύση, κάποιο κέντρο αποκατάστασης από ριζοσπαστικοποίησης ας πούμε σημαντικό είναι να υπάρχουν προγράμματα έγκαιρης απορριζοσπαστικοποίησης και να τα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι αρχές επιβολής του νόμου να έχουν τη δυνατότητα εγκαίρως να παρεμβαίνουν. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται ε, εντολή, εντολή που πρέπει εμείς να τη δώσουμε Αυτό όμως προϋποθέτει διάφορες ενέργειες. Προϋποθέτει να έχουμε τη δυνατότητα να συλλάβουμε κάποιον όπως την ε, περίπτωση του 29χρονου Βόρειο Αφρικανού που το προλάβαμε στο παραπέντε. Χρειάζεται και οι αρχές να έχουν κάποιο περιθώριο ελιγμών έτσι ώστε να μπορέσουν να συμπληρώσουν ε, το έργο των ε, δικαστικών αρχών. Όπως είπε και ο εισαγγελέα ε, Πιατσέντε, θέλουμε να διατηρηθεί η ελευθερία της μετακίνησης. Αλλά όταν κάποιος ταξιδεύει με τρομοκρατικές προθέσεις για να λάβει μέρος σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα στη Συρία ή να εκπαιδευτεί μόνος του ή δεν ξέρω και εγώ να πάει στη Συρία έτσι να εμπνευστεί, τότε πρέπει να είμαστε στη θέση να αντιδράσουμε και να αποτρέψουμε αυτούς τους ανθρώπους από το να διαπράξουν αδικήματα. Είναι πολύ δύσκολο έργο, δεν λέω ότι είναι εύκολο και δεν πρέπει να το ε, αντιμετωπίσουμε ε, με ελαφρότητα. Ο Άξελ πιστεύω πως είχε ε, δίκιο, παρότι πολλές φορές δεν συμφωνούμε και απόλυτα και ο Μίχαλ Μπόνι το είπε, χρειάζεται η συλλογή δεδομένων να είναι συλλογή σχετικών δεδομένων, χρήσιμων δεδομένων. Γι' αυτό και αυτά τα δεδομένα ε, πρέπει να ε, ανταλλάσσονται και αυτή η ανταλλαγή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, υποχρεωτική. Γι' αυτό στηρίζω αυτή την πρόταση 100%. Πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά και να είστε σίγουροι ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν κατέληξαν σε αυτές τις αποφάσεις τυχαία. Δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση. Και σίγουρα ε, αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες, όπως είπατε και εσείς, ναι, ε, παρουσιάστηκα στο Συνταγματικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στη χώρα μου και το δικαστήριο αποφάνθηκε ε, κατά αυτόν. Α, ε, γι αυτό, αυτό τι δείχνει. Δεν δείχνει ότι ήταν λάθο. Δείχνει ότι χρειάζεται ένα σαφέστερο ορισμό. Και ναι, να σα απαντήσω πριν προλάβετε να με ρωτήσετε, έχω διαβάσει όλη τη δικαστική απόφαση, ξέρω γιατί μιλάω. Αλλά όχι μόνο αυτό, βλέπω ότι κάποια συνταγματικά δικαστήρια ακριβώς εξαιτίας αυτής της απειλής που έχει ε, εμφανιστεί τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους παρομοίως και με το γερμανικό συνταγματικό ε, δικαστήριο κάποτε μπορούσαν να χαρακτηρίσουν αποφάσεις ως αντισυνταγματικές 100% τελεία και παύλα τώρα δεν είναι τόσο σπρώμαυρα τα πράγματα. Ο στόχος είναι να αποτρέψουν τους ε, τρομοκράτες να διαπράξουν σοβαρά εγκλήματα. Χρειάζεται όμως μια εξισορροπημένη διαδικασία με όλα τα πιθανά ε, μέτρα από το σοφρονισμό στις φυλακές, από τις προληπτικές δράσεις, από τα προγράμματα απορριζοσπαστικοποίηση. Χρειάζεται ένα συνδυασμό όλων αυτών και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε πολύ πιο έτοιμοι από ό,τι ήμασταν 25 χρόνια πριν. Τώρα, υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήξερα και τα έμαθα πρόσφατα ότι παρακολουθούνται αυτές οι ενέργειες ριζοσπαστικοποίησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2000, 2000 κάτι και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία ξέρετε δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Πέρασαν, πέρασε δεκαετία και βάλε μέχρι να οδηγηθούμε στο σημερινό σημείο, στη σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν θα μπορούσα να προτείνω, επειδή εσείς δεν έχετε ακούσει αυτά που ακούσαμε εμείς, να καλέσουμε εδώ σε αυτήν την Επιτροπή κάποιον εισαγγελέα, ε, κάποιον εμπειρογνώμονα, έτσι ώστε να ε, ακούσετε κι εσείς τι συμβαίνει τι έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές, πώς προσπαθούν να ε, υπερασπιστούν τα δικαιώματά μας και ταυτόχρονα να πιάσουν τους εγκληματίες. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα επιθυμούσα να είμαστε ενωμένοι στην αποφασή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ψηφίσουμε στις 24 Μαΐου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Θέσπιση μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ακολουθούμε διάφορα βήματα. Ετοιμάζουμε έγγραφα εργασία, ακρόασης, παρουσίαση ειδικών με μελέτη και τώρα έχουμε το σχέδιο έκθεσης. Η συγγήτρια λοιπόν η κυρία Σοφία Χετφέλτ παρακαλώ να μας παρουσιάσει αυτήν την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι σωστό η Επιτροπή μας Διακόπτη Πρόεδρος, παρακαλώ. Αν θέλετε να αποχωρήσετε από την αίθουσα, αποχωρήστε ησύχως, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, ησυχία στην αίθουσα. Ευχαριστώ, Σόφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, είναι σωστό στην Επιτροπή μας να μιλάμε και για το πώς θα ενισχύσουμε καλύτερα τις δικές μας αξίες. Μιλάμε πολύ για το πώς υποστηρίζουμε τις αξίες ε, αυτές στις επιθέσεις που δεχόμαστε απ' έξω. Στη διαδικασία θα θυμόσαστε ότι πρώτα είχαμε έγγραφα εργασίας, το οποίο επέβαλαν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και ο κύριος Σούφλιμ που ήταν υπεύθυνο συντάκτης νομοδότησης από την ΑΦΕΤ και εγώ έπρεπε όλα αυτά να τα συγκεράσω σε μία ενιαία έκθεση, μία πρόταση. Δεν ήταν εύκολο γιατί ακόμα και αν το άρθρο 2 μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά στη συνθήκη, τελικά δεν έχουμε κατάλληλη νομική βάση για να το θέσουμε σε εφαρμογή το άρθρο αυτό. Οπότε έψαξα δεξιά-αριστερά σε όλα τα έγγραφα εργασίας. Χρησιμοποίησα διάφορες μελέτες ειδικών και πυρογνωμόνων και τις μελέτες που ζήτησε η ίδια η Λίμπε, το έγγραφο της ΦΡΑ και κάποιες άλλες μελέτες. Υπογραμμίζω εδώ ότι υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες ε, γραμμές που χρησιμοποίησα σαν αρχές. Η πρώτη αρχή είναι ότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια πρώτη πρόταση και όσον αφορά εμένα τουλάχιστον είναι το σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας. Δεν λέω ότι το κείμενο αυτό θα μας οδηγήσει μέχρι το τέλος της διαδικασίας χωρίς να αλλάξουμε ούτε κόμμα. Όχι. Δεύτερη αρχή. Ό,τι μηχανισμό και αν τελικά αποφασίσουμε πρέπει να είναι αντικειμενικός ουδέτερος και να εφαρμόζεται εξίσου σε όλες τις χώρες μέλη ώστε η διαδικασία να αποπολιτικοποιηθεί. Έπειτα, δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, άρα τον νέο μηχανισμό πρέπει να το χτίσουμε πάνω σε ήδη υπάρχοντα μέσα όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Έχουμε ήδη ένα πλαίσιο κρατούς δικαίου, έχουμε ε, το διάλογο του Συμβουλίου και έχουμε ένα σωρό άλλα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Είπα ότι πρόκειται για τη διαδικασία εδώ. Δεν είναι μια απόφαση, μια και έξω, που δεν αλλάζει. Δεν βάζουμε εδώ προδιαγραφές. Είναι μια διαδικασία που προχωρά και ακόμα και αν αποφασίσουμε για ένα μηχανισμό, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να εμπλουτιστεί, να αλλάξει, να τροποποιηθεί ενδεχομένω τα επόμενα χρόνια. Γιατί μπορεί οι βασικέ αρχέ να παραμείνουν ίδιε, ο τρόπο με τον οποίο τι βλέπουμε στον κόσμο αλλάζει με τι εποχέ. Δεν πρέπει να είναι μια στατική απόφαση. Μια άλλη σημαντική αρχή είναι ότι θέλω ένα μηχανισμό που να μην απορρέει από μια κρίση. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αν θα εφαρμόζουμε ναι ή όχι το άρθρο 7, είναι θα εφαρμόζουμε ναι ή όχι άλλες κυρώσεις εναντίον της μιας ή της άλλης χώρας, γιατί τότε καταλήγουμε να βάζουμε τη μία χώρα σε αντιπαράθεση με όλους τις υπόλοιπες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι καρποφόρο. Προτιμάμε ένα μηχανισμό που να προβλέπει μόνιμο έλεγχο όλων των χωρών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρέπει να είναι μια διαδικασία η οποία ενισχύει την οτροπία του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και που αποτρέπει παραβιάσεις των αρχών αυτών και οδηγεί σε αποκλιμάκωση. Δεν περιλαμβάνει διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις. Αν αυτά υπάρχουν πρέπει να βασίζονται σε αποδείξεις. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν. Προσπαθούσα να βρω την κατάλληλη νομική βάση για ένα τέτοιο μηχανισμό και δεν ήταν εύκολο, όπως είπα. Δεν υπήρχε μία νομική βάση που να μας προσφέρει όλες τις επιλογές που θέλουμε. Επέλεξα τελικά τη διαθεσμική διοργανική συμφωνία. Δεν είναι με καλύτερη λύση, αλλά είναι ρεαλιστική, αν μη τι άλλο. Τίμασα, λοιπόν ένα σχέδιο διοργανικής συμφωνίας ως παράτημα στην έκθεσή μου που περιλαμβάνει τα εξή. Πρώτον, DRF βαθμολόγιο, δηλαδή δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα. Ένα βαθμολόγιο για αυτά τα τρία. Με ειδικέ αναχώρα εκθέσεις από πάνελ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Το δεύτερο είναι το εξάμεινο με κοινοβουλευτική συζήτηση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια με διευθετήσεις για την ε, αποτροπή διόρθωση βάση του 7. Και τέλος, ο κύκλος DRF, δηλαδή πάλι Δημοκρατία Κρατος Δικαίου και Θεμελιώδη Δικαιώματα. Γιατί, εντάξει, αξιολογούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να δούμε και εμείς κατά πόσο τηρούμε τις προδιαγραφές που θέτουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, άρθρο προς άρθρο. Πάντως χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που ήδη υπάρχουν. Και έχουμε πάρα πολλά εργαλεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το βαθμολόγιο για τη δικαιοσύνη, το CVM, για την Βουλγαρία και την Ρουμανία. Έχουμε τις εκθέσεις για τη διαφθορά, έχουμε για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και για τις ε, και άλλα εργαλεία για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ένα νέο σύστημα με ένα βαθμολόγιο και ειδικέ αναχώρα εκθέσεις. Αυτά τα δύο θα αποτελούν τη βάση για συζήτηση που θα γίνεται ετησίω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και τελικά, αν χρειάζεται, θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε μια προσέγγιση βήμα-βήμα προς το άρθρο 7, εάν χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ελπίζω ότι ο μηχανισμός θα φτάνει και θα είναι περιττό το να προσφεύγουμε στο άρθρο 7. Τέλος. Το κλειδί για όλα αυτά είναι η εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό και επέλεξα μια προσέγγιση η οποία ελπίζω θα καταλάβετε ότι απορρέει από την συνένεση. Συνένεση θέλω. Δεν θέλω τροπολογίες και πλειοψηφία με 51% γιατί αυτό δεν φτάνει. Δεν πρέπει να το δούμε σαν κάτι που επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις ε, των πολιτών, της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, όλων εδώ. Γι' αυτό και έκανε την προσπάθεια να έρθω σε επαφή με το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα Εθνικά Κοινοβούλια, για να πετύχουμε συνένεση. Η διαδικασία αυτή είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Τέλος, υπάρχει σχέδιο χρονομοδότησης της ΑΦΚΟ. Υπάρχουν και τροπολογίες θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε. Συνέχεια μου έρχονται ειδοποίησεις από ανθρώπου που ενδιαφέρονται και εγώ ανάλογα με τα σχόλια που θα έχω ακούσει θα υποβάλω τροπολογίες και θα οργανώσω και διάφορα γεύματα, Ήδη είχα δύο μέχρι τώρα. Δεν πρόκειται για μεγάλα γεγονότα, αλλά αν ευρωβουλευτέ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να μα το πούν με μη κυβερνητικέ οργανώσει, με δικαστικά σώματα, διεθνείς οργανισμούς, υπαλλήλου, οργανώσεις καταναλωτών, θρησκευτικέ και μη θρησκευτικέ οργανώσεις, σύλλογοι δημοσιογράφων. Η προθεσμία θα είναι η 13η Μαΐου για την υποβολή τροπολογιών. Και η πρώτη συζήτηση θα γίνει νομίζω 21 Μαΐου, ούτε σπάω κάτι τέτοιο. Προσβλέπω λοιπόν στα σχόλιά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να ακούσουμε τον για την κυρία Άγγελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου ζήτησε ο Φρανκ να τον εκπροσωπήσω σήμερα και να παρουσιάσω τις απόψεις του και να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί θα χρειαστεί να φύγω αφού παρουσιάσω τα σχόλια του κυρίου Άγγελ γιατί πρέπει να πάω στο αεροδρόμιο. Κατά την άποψη του Φρανκ συνάδει το σχέδιο έκθεσης με όλες τις συζητήσεις, με όλους τους σκιώδες. Ε, ε, κυριάρχησε επικοδομητική ατμόσφαιρα σε όλα τα βήματα. Αποσκοπεί δύναμη του άρθρου 292 να δημιουργηθεί μια συνθήκη για δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, υπό τη μορφή διοργανικής συμφωνίας που θα ορίζει τις διευθετήσεις που θα διευκολύνουν τη συνεργασία των θεσμών και των κρατών μελών στο πλαίσιο του άρθρου 7 της Συνθήκης Λειτουργίας θα περιλαμβάνει τους ε, υπάρχοντες μηχανισμούς και τις πρακτικές. Ο Φρανκ θεωρεί ότι το άρθρο 295 είναι η μόνη διαθέσιμη νομική βάση για το σύμφωνο και η μορφή διοργανικής συμφωνίας είναι η μόνη που μπορεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα και των τριών θεσμών στον τομέα. θα βασίζεται σε μια λογική όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού Πολιτικής. Θα συμπεριλαμβάνει μια γενική αξιολόγηση του ιστορικού και των αποτελεσμάτων κάθε κράτους μέλους ετησίως και έναν κύκλο κοινοβουλευτικής συζήτησης και στο Ευρωκοινοβούλιο βάσει των συστάσεων κατά χώρα. Με τον τρόπο αυτό ο μηχανισμός δεν θα χρησιμοποιείται κατά περίπτωση. Κάθε φορά προκύπτει κάποιο ζήτημα σε ένα κράτος μέλος θα είναι ένα μόνιμο εργαλείο αξιολόγησης όλων των κρατών μελών κάθε χρόνο, ώστε να προσδιορίζεται κατά πόσο παρατηρούνται αποκλήσει από ορισμένα πρότυπα στους τομείς που αναφέρουμε. Ο μηχανισμός βασίζεται σε ένα βαθμολόγιο που θα ε, καταρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και θα έχει οθετηθεί από την Κομισιόν. Παρότι η οθέτηση από την Κομισιόν φαίνεται λογική διότι είναι θεματοφύλακα των συνθηκών και υπάρχουν διατάξεις στον τομέα, ε, η ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, δημιουργεί πρόβλημα. Το μέγεθο, η σύνθεση και με ποια λογική θα επιλέγονται τα μέλη μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Οπότε δεν έχουμε ενδείξει βέβαια ότι δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια ο πάνελ. Το ζήτημα είναι με ποια μορφή και πώ θα ορίζεται. Αν παρουσιαστούν προβλήματα θα υπάρχει μια αυτόματη προσφυγή στο άρθρο 7 και αυτό θέτει δύο ερωτήματα. Το πρώτο, το άρθρο 7 ξαφνικά θα τεθεί σε εφαρμογή, θα ενεργοποιηθεί εδώ και καιρό. Περιγραφτεί ως ένα άρθρο με αμφίβολο περιεχόμενο και στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει να χάσει δικαιώματα ψήφου ένα κράτος ο Φρανκ λέει ότι αυτό δεν έχει κάτι σκληροπυρηνικό. Είναι πολύ λογικό η συνθήκη με την οποία έχουν δεσμευτεί όλα τα κράτη-μέλη να βασίζεται σε συγκεκριμένε αρχέ και να τηρείται από τα κράτη-μέλη. Και αν δεν τηρείται, να υπάρχει κάποια ε, κάποιο αποτέλεσμα γι' αυτό. Ένα κράτος, ε, οποιοδήποτε κράτος υποχρεούται να τηρεί τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την προσχώρηση, αυτά είναι τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. Αφού βρίσκεται εντό τη Ένωση, δεν μπορεί να επιτρέπεται να παραβιάζει τα πρότυπα αυτά χωρίς συνέπειε. Η δεύτερη ερώτηση. Η χειρότερη, ε, το χειρότερο αποτέλεσμα θα ήταν η απώλεια δικαιωμάτων ψήφου. εάν κάποια χώρα οδηγείται σε δικτατορικό καθεστώς ε, ε, το άρθρο 7 είναι αρκετό το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να παραμείνει μέλος αν το επιθυμεί το ερώτημα λοιπόν είναι το άρθρο 7 λύνει το πρόβλημα αυτό ε, όλα αυτά επικεντρώνονται στο εξή επιχείρημα μπορεί να χρειαστεί αλλαγή των συνθήκων για όλο αυτό αυτό θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε στο τελικό κείμενο που θα συμφωνήσουμε ωστόσο. Το άρθρο 295 φαίνεται να είναι η επαρκή βάση για την υιοθέτηση της παρούσας έκθεσης και για την ε, σύνταξη μιας διοργανικής συμφωνίας στον τομέα. Ρόμπερτα, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που αντικαταστήσατε τον Φρανκ. Το λόγο έχει η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει σε ένα τόσο δύσκολο θέμα και για τις διαβουλεύσεις που ήταν πραγματικά εύρυες. Εκτίμησα ιδιαίτερα την προσπάθεια να βρεθεί η κατάλληλη νομική βάση η οποία να επιτρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια των συνθήκων και τα όρια των συνθήκων ώστε να καθορίσουμε ένα εργαλείο το οποίο να μπορέσει να λειτουργήσει σύντομα χωρίς να απαιτεί ε, αναθεώρηση άμεσα των συνθήκων. Τα παρομοίως θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσες και συμφωνώ με αυτές με τις προτάσεις που υπάρχουν στην έκθεση. Αναφέρομαι στην ιδέα δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου νομικής αρρωγής προς τους πολίτες σε περίπτωση διαδικασιών ε, για παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Συμφωνώ και με τις προτάσεις ε, ε, υποθετικής αναθεώρησης ε, των συνθήκων. Σκεφτούμε στην την κατάργηση του άρθρου 51 ε, του χάρτη και για το άρθρο 2. Τη δυνατότητα δηλαδή των πολιτών να ε, καταφυγούν στο δικαστήριο. Όσον αφορά τον επίκεντρο της δουλειάς αυτής, δηλαδή που είναι η διοργανική συμφωνία, θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις. Είναι σημαντικό το τμήμα 1 του εγγράφου ε, για το βαθμολόγιο. Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόταση ε, του να υπάρχουν πολλές διαφορετικές ε, απόψεις αξιόπιστες παρότι μου φαίνεται υψηλό ο αριθμό των εμπειρογνωμών που αναφέρεται. Επίση, εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών συγκεκριμένων βασισμένων στι σημερινέ εξελίξει ε, στον τομέα των δικαιωμάτων και του κρατού δικαίου και στο γεγονό ότι η άποψη των εμπειρογνωμών θα αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων. Και επίση, εκτιμώ την πρόταση ε, διασφάλισης της αυτονομίας του οργάνου αξιολόγησης. Θα ήθελα εδώ όμω να αναφέρω κάποιες επιφυλάξει για τρία σημεία. Πρώτον, το follow-up ε, και το βαθμολόγιο. Κεντρικό ρόλο όσον αφορά την αξιολόγηση αυτού αναλαμβάνει το Συμβούλιο μέσω του μέσου ετησίου διαλόγου. Δεν συμφωνώ απόλυτα με την ιδέα του να αναθέσουμε τον έλεγχο της συμπεριφοράς των ε, κρατών στο όργανο που τα εκπροσωπεί. Καλύτερα ίσως ένα ανεξάρτητο όργανο. Ταυτόχρονα ε, έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων. Η ενοποίηση των σημερινών ε, εργαλείων σύμφωνα, σίγουρα επιτρέπει να αποφύγουμε τη δύσκολη αναθεώρηση των συνθήκων, αλλά ταυτόχρονα επί της ουσίας δεν αλλάζει τη σημερινή κατάσταση που βασίζεται ε, στην προσφυγή στο άρθρο 7, το οποίο ε, παρουσιάζει κάποια πολιτική ευαισθησία και ε, που γίνεται απουσία παρέμβασης του δικαστηρίου. Δεύτερον, η ανάλυση και η παρακολούθηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης όταν παραβιάζουν δικαιώματα και κράτη δικαίου και το κράτος δικαίου, συγγνώμη. Η εκθέση λέει καθαρά ότι ο υπεξέταση μηχανισμό θα πρέπει να εφαρμόζεται είτε στα κράτη-μέλη είτε στα θεσμικά όργανα. Εξίσου και στα δύο. Αυτή η πρόταση διοργανική συμφωνία, ωστόσο, τελικά δημιουργεί ένα διπλό σύστημα στο οποίο σε τελική ανάλυση το βαθμολόγιο δεν εφαρμόζεται ε, για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπροσθέτως, ε, η διοργανική συμφωνία φαίνεται να δεσμεύει μόνο τις, ε, τα υπογράφοντα όργανα, εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογή μια σειρά οργάνων, οργανισμών πολύ σημαντικών της Ένωσης. Κατά την άποψή μου, για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός ο μηχανισμός για την προστασία του κράτους δικαίου και των ε, δικαιωμάτων και της δημοκρατίας πρέπει να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φάσμα ε, οργανισμών και θεσμών όλων όσων λειτουργούν υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να γίνεται μια ρητή αναφορά στα θεσμικά οργάνα όπως το Συμβούλιο φυσικά και η Κεντρική Τράπεζα αλλά και σε άλλους οργανισμούς όπως η Ευρωπόλ αλλά και σε άτυπου οργανισμούς όπως το Eurogroup που ενδέχεται να παραβιάσουν θεμελιώδη δικαιώματα. Η ανάλυση της αγωγής ε, των ε, διαφορών οργανισμών μπορεί να αποτελέσει παράμετρο αξιολόγησης της λειτουργίας ελέγχου και επίβλεψης που θα ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά την άποψή μου, είναι επίσης σημαντικό να πάμε πιο πέρα από την αξιολόγηση της καθαρά νομοθετικής φάσης και να λάβουμε υπόψη όλες τις πράξεις που δυνάμει του άρθρου 263 μπορεί να έχουν νομικά αποτελέσματα ενώπιον τρίτων. Τρίτο και τελευταίο σημείο, τα κοινωνικά δικαιώματα. Το scoreboard, το βαθμολόγιο, εισάγει ρητά τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων ως δίκτυ επιδόσεων. Ωστόσο, μια τέτοια ανάλυση θα περιοριζόταν από τις διατάξεις του ίδιου του χάρτη που ορίζουν την εμβέλεια των κοινωνικών δικαιωμάτων που ονομάζονται αρχές στο χάρτη που είναι λιγότερο πιο αδύναμα από τα ε, πολιτικά δικαιώματα. Κατά την άποψή μου καλό θα ήταν η αξιολόγηση να συμπληρώνεται και με άλλα κριτήρια. Στο μέλλον μάλιστα θα πρέπει να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο προσχώρησης της Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη ώστε να συμπεριληφθεί ο χάρτης αυτός, ο κοινωνικός χάρτης, σε αυτό που ορίζουμε ως ε, διαδικασία, ε, ώστε αυτή την έκθεση εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λούνατσεκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως ε, μπορώ να είμαι σύντομη, διότι έτσι όπως παρουσίασε η Σοφία Ιντφέλντ τα ε, διάφορα θέματα, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι ε, δείχνουν ότι έχουμε τις ίδιες απόψεις. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Σοφία Ιντφέλντ την προσέγγιση που υιοθέτησε. Είναι μια προσέγγιση που ε, προσπαθεί να παρουσιάσει ένα μοντέλο ένα μηχανισμό που θέλει να συνδυάσει τον διάλογο με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, δημιουργώντας έτσι αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μια εμπιστοσύνη που έχει χαθεί, έχει χαθεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Ένας μηχανισμός όπως τον παρουσιάσατε, μια διοργανική συμφωνία, η οποία σε είναι κάτι που ζητούσαμε συνεχώς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια τακτική αναθεώρηση και ε, έλεγχος κάθε κράτους μέλους έτσι ώστε να μην ε, υπάρχει εντύπωση ότι οι κακές Βρυξέλλες είναι πάνω από τα κεφάλια τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρω πως είναι σημαντικό διότι όπως γνωρίζετε είμαι από την Αυστρία και το 2000 είχαμε τις... Ε, λεγόμενες κυρώσεις ε, κατά της ε, δεξιάς λαϊκιστική κυβέρνηση. Εγώ ήμουν στην αντιπολίτευση τότε και ήμασταν υπέρ αυτών των κυρώσεων, οι οποίες στην ουσία δεν ήταν κυρώσει, διότι δεν υπήρχε μηχανισμός κυρώσεων. Καταρχάς δεν υπήρχε στρατηγική εξόδου. Πάντα όταν ε, χαράσεις μια στρατηγική πρέπει να έχεις και μια ε, ασφαλιστική δικλίδα για να ε, Φύγει από αυτή τη στρατηγική. Τώρα, Ουγγαρία, Πολωνία και άλλα κρατημέλη έχουν βρεθεί στην ίδια θέση και όλοι λένε ότι οι Βρυξέλλες μας τα κάνουν αυτά και χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα, στο εμείς και στο αυτοί. Αυτό δεν ισχύει όμως, δεν είναι εκείνη εναντίον των άλλων. Πιστεύω λοιπόν πως με μια τακτική αναθεώρηση, τακτικό έλεγχο όλων των κρατών μελών θα βελτιωθεί η κατάσταση, διότι κανείς δεν είναι τέλειος. Είναι ένα αρκετά καινοτόμο μοντέλο και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο και με τα άλλα θεσμικά όργανα θα δημιουργήσουμε κάτι που θα χτίσει περισσότερη εμπιστοσύνη και θα βγούμε από αυτό το τέλμα ε, της ε, αδράνειας. Αυτό το άρθρο 7 Αυτό λοιπόν ε, είναι κάτι που η πολιτική μου ομάδα στηρίζει απόλυτα και πιστεύω πως η Σοφή είχε την ιδέα να καλέσει διάφορους φορείς από πολλά επίπεδα για ανταλλαγή απόψεων. Είναι ένα πάρα πολύ ε, καλό στοιχείο, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Πιστεύω πως η πλειοψηφία είναι μαζί σου. Γι' αυτό πιστεύω πως αυτή η νέα Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων είναι καλή ιδέα. Ορισμένοι εξέφρασαν την κριτική τους για το μέγεθος της Επιτροπής. Λένε ότι είναι πολύ μεγάλη, όμως δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σίγουρα καταλαβαίνω το γεγονός ότι κάποιοι θα θεωρούν ότι υποεκπροσωπούνται ή ότι δεν εκπροσωπούνται, αλλά πιστεύω πως είναι μια καλή αρχή και θα δούμε εάν στη συνέχεια θα είναι αρκετός αριθμός των συμμετεχόντων και ε, το εύρος που θα έχει. Πιστεύω πως είναι μια καλή αρχή και θα μπορέσουμε μετά στη συνέχεια να μπούμε σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό στηρίζω και τη στρατηγική και το περιεχόμενο παρά τα μικρά λαθάκια τεχνικής φύσεως που θα μπορούμε να λύσουμε, είμαι σίγουρη. Επίσης, ε, Σίγουρα μια αλλαγή στις συνθήκες είναι κάτι ε, τολμηρό που θα μας φέρει παραπέρα, όμως δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως η αρχή είναι καλή, θα καταφέρουμε να έχουμε με το πλευρό μας αρκετούς. Ελπίζω και το Συμβούλιο και την Επιτροπή και την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Αλλά αυτά που άκουσα μου δημιουργούν αισιοδοξία. Είναι όντως μια καλή αρχή. Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το άρθρο 7 λέει αυτά που λέει όχι τυχαία. Και ούτε είναι τυχαία που δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εύκολα. Όντως δεν συντάχθηκε ώστε να χρησιμοποιείται. Ακούμε ότι ζούμε σε δημοκρατικές χώρες και ότι μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για καμία χώρα μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη δημοκρατία σε κάποια χώρα μέλους. Το άρθρο αυτό όμως δεν έχει συνταχθεί για να ελέγχεται επιμονή μου βάσεως κανείς. Και μιλάει για κυβερνήσεις, για χώρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν μπορεί να αναλάβει δράση βάσει του άρθρου 7. Και όταν ακούσαμε πρόσφατα συζήτηση για την Πολωνία, δεν είχαμε απάντηση για νομική βάση που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για την Πολωνία. Και αυτό γιατί ο νόμος λέει ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια αμφιβολία για την κατάσταση σε οποιαδήποτε χώρα, τότε το αναθέτει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα. Οπότε η προσπάθεια δημιουργίας νέου μηχανισμού αντιβαίνει στη συνθήκη όσο έχει τώρα. Και θα ήταν μια διαφορετική η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτήν στην οποία προσχωρήσαμε εμείς. Η συζήτηση λοιπόν για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ναι, είναι απόλυτο θεμητή. Μπορούμε να συζητήσουμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Και εγώ έχω τις δικές μου ιδέες για τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στην Ολλανδία. Το δικαίωμα το δίκαιο δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί σύμφωνα με, την, με τόσα προτείνεται. Κανείς δεν μπορεί όμως να ζητήσει από το κράτος να βοηθήσει κάποιο άτομο να παρετηθεί από τα δικαιώματά του. Και αυτό ακριβώς είναι η νομική βάση της Πολωνίας. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν μ' αρέσει επίσης ούτε και ο τρόπος με τον οποίο έγινε το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για τα ομοφιλοφιλικά ζευγάρια. Και εδώ έχω εγώ αμφιβολίες όσον αφορά την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Γιατί η Ιρλανδική νομοθεσία δεν δίνει την δικαιότητα, ε, το δικαίωμα, συγγνώμη, δεν δίνει το δικαίωμα να οργανώνονται δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία που λαμβάνεται σε άλλη χώρα. Το σύστημα λοιπόν στην η Ιρλανδία, ναι μεν έχει αναπτυχθεί πολύ, αλλά θα έπρεπε όλες οι πλευρές να έχουν δικαίωμα στα μέσα ενημέρωσης. Δεν έγινε όμως αυτό. Στο Κοινοβούλιο μπορούμε να συζητάμε, μπορούμε να ταξιδεύουμε, να πηγαίνουμε σε άλλες χώρες, να υπάρχει διάλογος, αλλά ο έλεγχος που προτείνεται αφορά μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι αυτή στην οποία ζούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να υπάρχει αλληλοβοήθεια μεταξύ των χωρών μελών, για να δημιουργηθεί μια αγορά η οποία να είναι συμβατή με τι τάσει που επικρατούν στο σύγχρονο κόσμο. Χρειαζόμαστε ολοκλήρωση των αγορών, χρειαζόμαστε τη στήριξη την πολιτική ο ένα του άλλου και στήριξη των χωρών που την έχουν ανάγκη, αλλά πρέπει να βοηθάει μια χώρα την άλλη, όχι να ελέγχει μια χώρα την άλλη. Δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ακόμα αν η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ήταν αρκετά αμερόληπτη για να αποφασίσει, μπορεί να είχε παρέμβει στη δημιουργία του και την οργάνωση του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Μην ξεχνάμε τα, τη γνωστή ρίση ότι μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα αγωνιστώ και θα δώσω την ίδια μου τη ζωή για να έχεις το δικαίωμα να υποστηρίζεις τις απόψεις σου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δημιουργήθηκε για να προωθεί τις εξελίξεις και για να βοηθάει όποιον χρειάζεται προστασία. Ή που είμαστε κοινότητα που βασίζεται σε αυτή την αρχή της αλλοβοήθειας ή αλλιώς δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μια εντελώ διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, εκτιμώ την προσπάθεια που έγινε για να ετοιμαστεί η πρόταση αυτή, αλλά εγώ πιστεύω ότι πάει προς την λάθος κατεύθυνση. Θέτει υποφυσβήτηση τη συνθήκη ή αλλιώς η συζήτηση που κάνουμε δεν έχει νόημα. Ο μηχανισμός αυτός βάσει του άρθρου 7 δεν μπορεί να αλλάξει. Ή λοιπόν που ζούμε σε έναν ουτοπικό κόσμο ή θέλουμε να παρακάμψουμε τον νόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπόνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα εστιαστώ στην πρόταση που παρουσίασε η Σοφίν Βέλτ και η Σκιώδης, αλλά δεν θα κάνω γενικές δηλώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Θεωρώ ότι αξίζει την υποστήριξή μας. Χρειαζόμαστε ένα σαφή μηχανισμό για το θέμα αυτό. Και το σύμφωνο που αναφέρεται στην πρόταση χρειάζεται ως εργαλείο για τη μελλοντική δεσμευσή των ενδιαφερομένων και των εταίρων και ως υποβαθρό για να λειτουργούν σωστά οι μηχανισμοί βάσει και της διοργανικής συμφωνίας. Ναι, έχετε δίκιο. πρέπει να είναι το αποτέλεσμα συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων, ώστε όλοι να εμπλέκονται στην ε, ε, υλοποίησή του. Πώ θα λειτουργήσουν ορισμένοι μηχανισμοί, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Για παράδειγμα, το ποιο θα πρέπει να συμμετέχει στο πάνελ εμπειρογνωμόνων, πώ αυτοί θα ορίζονται και τι αρμοδιότητε και τι γνώση θα πρέπει να έχουν. Αλλά επίση και τι είδου νομικέ γνώσει θα έχει το πάνελ και τι ρόλο θα παίζουν οι συστάσει του πάνελ, για παράδειγμα αλλά είμαι υπέρ της ε, εφαρμογής ε, της δημιουργίας αυτού του πάνελ. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε σαφώς επιλεγμένους δείκτες που να ε, εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη εξίσου. Και φυσικά όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι διατεθειμένα να ανταλλάξουν απόψει. Αυτό που είναι σημαντικό και σαφές για μένα είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ποσοτικοί δείκτες αλλά και ποιοτικοί. Ωστόσο πρέπει να διασφαλίσουμε την αντικειμενικότητά τους. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην βλέπουμε μόνο αριθμού στις αξιολογήσεις μας. Συμφωνώ ότι αυτό ο μηχανισμό γενικότερα θα πρέπει να είναι κάτι ζωντανό. Θα πρέπει να γίνει μετά από διαβούλευση με τα κρατικά κοινοβούλια. Η φωνή του πρέπει να ακουστεί σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρω ότι η συζήτηση αυτή μπορεί να μην φαίνεται αρκετή για πολλούς από εμά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει κάποια αξία από μόνη τη Θα μπορούσε να επηρεάσει πολύ σημαντικά το επίπεδο ε, συμμετοχής στη δημοκρατία. Η δημοκρατική συμμετοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να την ξεχνάμε όταν ε, συζητάμε αυτή την έκθεση. Για παράδειγμα, ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση αυτής της συμμετοχής καθιστώντα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων πιο διαφανή, επιτρέποντα ευρύτερη διαβούλευση με τους οργανισμούς μεν, αλλά και με ανθρώπους χρησιμοποιώντας τις μορφές του crowdsourcing ε, για να λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μην ξεχνάμε ότι οι πολίτες μας αποτελούν για μας πηγή γνώσης, ε, για μας για τις δημόσιες αρχές και ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στον κοινωνικό και δημοκρατικό διάλογο στον οποίο δεν θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο ε, υπάλληλοι ε, και οι διεθνείς οργανισμοί χρειαζόμαστε και την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους τους ε, εκπροσώπους των πολιτών. Ε, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη, για τη σύνθεση του πάνελ. Με ενδιαφέρει λοιπόν πολύ αυτή η συζήτηση και ευχαριστούμε που την προτείνατε και επίσης θα πρέπει να δούμε το ρόλο του άρθρου 7 και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πραγματική ερμηνεία αυτού του άρθρου. Επειδή και εγώ είμαι Πολωνός, θα ήθελα να πω ότι Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Μαρέκ με το γεγονό ότι μπορεί να κάνει δήλωση δηλαδή, αλλά δεν ε, συμφωνώ με το περιεχόμενό τη. Ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ε, η συγκήτρια, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχολεία τους. Να απαντήσω στα γρήγορα σε διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στον κύριο Γιουρέκ. Ε, θα ήθελα να, να ξεκαθαρίσουμε δύο παρανοήσεις. Λέτε ότι το άρθρο 7 δεν είχε δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθεί. Ναι, πρακτικά έτσι φαίνεται να είναι. Ωστόσο, δεν πάμε να αποτελεί ένα άρθρο της συνθήκης. Και αν θεωρούμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να το διαγράψουμε. Αν δεν το διαγράψουμε, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλιώς είναι ανόητο να υπάρχει. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι το αντίθετο της προσπάθειας ελέγχου κάποιου. Διότι οι μηχανισμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή φαίνεται να προσπαθούν να ελέγξουν και να επιβάλλουν πράγματα. Αλλά ουσιαστικά η προσπάθεια που κάνουμε εδώ είναι το αντίθετο, να προσπαθήσουμε να έχουμε ανθρώπου με το μέρο μα και να κάνουμε αυτή την πραγματική δημόσια συζήτηση. Πάντα λέμε για κοινέ αξίε, μιλάμε για κοινέ αξίε. Αλλά δεν ξέρουμε ποιε είναι αυτέ. Ξέρουμε τα βασικά, εντάξει, όλα έχουν γραφτεί σε διάφορα έγγραφα, αλλά οι κοινέ αξίε είναι το αποτέλεσμα μια δημόσια συζήτηση ε, με συμμετοχή όλων, όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Επίσης ε, είπατε κάποια πράγματα για το πάνελ εμπειρογνωμόνων. Θα έπρεπε να είχα πει κάτι αυτό, γι' αυτό στην εισαγωγή μου. Ουσιαστικά το μόνο που προτείνω, ε, το πάνελ το μόνο νέο πράγμα προτείνω. Όλα τα υπόλοιπα βασίζονται σε υπάρχοντα μέσα και την εξέλιξη υπαρχόντων μέσων. Και ναι, και ο Ρίκη είχε δίκιο. Επίτηδες ε, προτείνω ένα τόσο ευρύ πάνελ διότι θα πρέπει ο κόσμος να εμπιστευτεί, να δείξει εμπιστοσύνη στη διαδικασία και για να αποδεχθεί το αποτέλεσμα. Εγώ εξέτασα διάφορα ενδεχόμενα, διάφορες επιλογές και με όλες τις άλλες επιλογές ο κόσμος μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται ότι αφήνουμε την Κομισιό να επιβάλλει καιρό σε χώρες και ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Οπότε χρειαζόμαστε ένα πάνελ το οποίο να φαίνεται αξιόπιστο στα μάτια όλων, ε, είναι αντιπροσωπευτικό και μπορούμε να συζητήσουμε Πολύ ωραία για το ποιο θα συμμετέχει σε αυτό, πώ θα ορίζονται κτλ. Εδώ εγώ έκανα μία πρόταση ουσιαστικά, έκανα μία λίστα και κατέληξα στον αριθμό του 66. 66 ε, μάλιστα είναι και το έτο που γεννήθηκα. Οπότε ίσως είναι συμβολικό αυτό, ίσως είναι ουράνια σήμα. Αλλά ε, εγώ το προτείνω και α δούμε τι άλλε ιδέε θα προτείνουν και οι υπόλοιποι. Κάποιες παρατηρήσεις ακούσαμε από την κυρία Σπινέλη πολύ ενδιαφέρουσες, ε, συμφωνώ με τις περισσότερες, αλλά μην ξεχνάτε ότι δεσμευόμαστε από το παρόν περιεχόμενο των συνθήκων όσον αφορά τις αρμοδιότητες και στη οποία εφαρμογή τη έκθεση, για παράδειγμα αυτό που λέτε για τα κοινωνικά δικαιώματα. Ναι, φυσικά η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να το διευρύνουμε πέραν του πεδίου του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά δεν είναι το θέμα αυτή τη έκθεση. Μπορεί να προκύψει τη διαδικασία με στα επόμενα χρόνια. Τέλος, για το άρθρο 7 ξανά, κατά πόσο θα ενεργοποιείται αυτόματα. Η ναι, κυρία Μέτσολα είπε όχι είναι η απάντηση. Όχι αυτόματα. Διότι αυτό απλά δεν είναι δυνατόν. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη συνθήκη. Το μόνο προσπαθώ να κάνω εδώ είναι να δημιουργήσω ένα μηχανισμό ο οποίο θα αποτελεί τη βάση. Γιατί όπω είπε πολύ σωστά ο κύριο Γιούρεκ, είπε ποια είναι η νομική βάση για μια τέτοια παρέμβαση. Γενικότερα, ποια είναι η βάση για οποιαδήποτε παρέμβαση. Εντάξει, μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε για ή να τσακωθούμε για την ε, νομική βάση, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουμε πιο συστηματικά, συγκρίσιμα μεταξύ κρατών μελών, ώστε να υπάρχουν κάποια πρότυπα που θα εξελιχθούν με το χρόνο και εκεί μπορεί πλέον να δημιουργηθεί μια βάση ενεργοποίηση του άρθρου 7 σε περίπτωση που κάποτε χρειαστεί κάτι τέτοιο. Αυτό πιστεύω ότι θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα τη όλη διαδικασίας και όπως είπε και ο κύριος Μπόνι να την κάνει πιο διαφανή. Πριν κλείσω να πω ότι την πρόταση αυτή εγώ την υποβάλλω ενώπιόν σας ε, και από τότε που την υπέβαλα έλαβα διάφορες νέες συστάσεις και προτάσεις που θα με οδηγήσουν να κάνω και εγώ τροπολογίες στη δική μου έκθεση. Ελπίζω να καταφέρουμε να την εμπλουτίσουμε στη διάρκεια της διαδικασίας και να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα τύχει ευρεία υποστήριξη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε, Σόφη. Τώρα, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Ερώτηση στην Επιτροπή του Ζωράρ Ντεπρέ σχετικά με τον αριθμό των κρατών μελών που θεωρούν την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2016 επεστάλλει ερώτηση και βάσει το 135 θα έπρεπε να είχε απαντηθεί σε 6 εβδομάδες η ερώτηση αυτή. Δεν απαντήθηκε όμως από την Επιτροπή μέσα στην προθεσμία. Κύριε Ντεπρέ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξηγήσατε με δύο λόγια το αντικείμενο του ζητήματος. Ρώτησα την Επιτροπή να μου πει ποιος είναι ο αριθμός των κρατών μελών που θεωρούν την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα. Διότι η συνέπεια εφαρμογής της ε, αρχής αυτής για μια χώρα στην πράξη έχει τεράστιε επιπτώσεις όσον αφορά του ετούντε άσυλο, γιατί αν έχω καταλάβει καλά, κάθε τον άσυλο, ο οποίος έχει περάσει τράνζιτ από μια χώρα η οποία θεωρείται ασφαλής, από μια χώρα μέλο, τότε δεν εξετάζεται η αίτηση επί τη ουσία από το κράτος μέλο, αλλά το άτομο αυτό επιστρέφεται στη χώρα τράνσιτ που θεωρείται ασφαλή. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία αυτό. Εξού και ερώτησή μου, πόσε χώρε μέλη θεωρούν ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα. Και κάτι ακόμα που δεν το επέβαλα στην ερώτησή μου, αλλά ρωτάω τώρα, η Επιτροπή μας έχει στείλει πρόταση με κατάλογο χωρών ασφαλών. Δεν σημαίνει βέβαια το ίδιο, αυτό σημαίνει ότι οι απάτριδες και οι υπήκοοι θα εξαρτιόνται από την απάντηση αυτή. Θέλω λοιπόν να ξέρω. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ για την απάντηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Έχει να κάνει με εσωτερικές διαδικασίες. Είναι στο δρόμο η απάντηση. Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, για το πλαίσιο. Εφαρμόζοντας την αρχή αυτή της ασφαλούς χώρας, οι χώρες μέλη μπορούν να ορίσουν ότι στο διεθνές δίκαιο μια και έξω η χώρα αυτή και για πάντα είναι ασφαλής. Αλλά μπορούν ανταυτού να εφαρμόσουν την αρχή που είναι κατά περίπτωση. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να περάσει την εθνική νομοθεσία σαν κάτι οριστικό. Τώρα, οι χώρες δεν έχουν ορίσει έτσι ως ασφαλή χώρα για πάντα την Τουρκία. Κατά το παρελθόν όμως και κατά περίπτωση από κάποιες χώρες μέλη μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Δεν το αποκλείω. Πάντως προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει σε, τέτοιο, σε τέτοια απόδοση καμία χώρα. Τώρα, κατά τα άλλα, εμείς δεν θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει τέτοια πρόταση με κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών. Αλλά μία διάταξη του κεκτημένου όταν θα περάσουμε στην αναθεώρηση για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε με πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις ασφαλείς τρίτες χώρε. ενδεχομένω θα το λάβουμε υπόψη μα αυτό. Ο κύριο Δεπρέ. Αν ήταν τόσο απλή απάντηση, δεν θα χρειαζόταν έξι εβδομάδε για να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τέλο πάντων, πλάκα κάνω. Λοιπόν, κατάλαβα καλά τι είπατε. Λέτε ότι για να σταλεί ένας ε, ετών άσυλο σε μια τρίτη χώρα, μπορούμε κατά περίπτωση να αποφασίσουμε ότι αυτή η χώρα είναι ασφαλής ή δεν είναι ακόμη και αν δεν έχουμε νομική βάση να το κάνουμε αυτό. Κατά περίπτωση το αποφασίζουμε. Λέτε, και θα επανέλθω στην ερώτησή μου, λέτε καμία χώρα μέλος δεν εφαρμόζει την αρχή της τρίτης χώρας. Η Ελλάδα δεν πήρε μια τέτοια απόφαση για να θεωρήσει ότι η Τουρκία είναι ασφαλής τρίτη χώρα. Η κυρία Ινθετφέλτ. Τελειώσατε. Μπορώ να επανέλθω μετά, Πρόεδρε. Ωραία. Η κυρία Χετφέλτ. Μα αν λέτε ότι η απόφαση για το κατά πόσο είναι ασφαλής μια χώρα ή όχι ή είναι κατά περίπτωση, μα αυτή είναι η τακτική διαδικασία για τις αιτήσει ασύλου. Και δεν είναι αυτή η έννοια της ασφαλούς χώρας. Εννοείται ότι η έννοια ο ορισμός μιας χώρας ως ασφαλούς δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν ατομικά να υποβάλουν τις αιτήσει ασύλου τους οι άνθρωποι. Το ότι απορρίφθηκαν κάποιες επειδή το συγκεκριμένο άτομο ε, θεωρήθηκε ότι δεν κινδυνεύει, δεν σημαίνει ότι θεωρείται και ασφαλής η χώρα από την οποία έρχεται. Ο κύριος Ντεπρέ να συνεχίσω μετά από αυτό που είπε η Σόφη. Θυμάμαι τις επιπτώσεις του ορισμού μιας χώρας ως ασφαλούς χώρας. Ότι τότε το αίτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί απαράδεκτο το αίτημα ασύλου, υποθέτουμε, ο κύριος Δεπρέ. Όλες οι αιτήσει ασύλου που διατυπώνονται λοιπόν σε μια τέτοια χώρα θεωρούνται απαράδεκτες, σωστά. Βάσει των όσων συμβαίνουν ε, σήμερα η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να υιοθετήσει αυτόν τον ορισμό για να κάνει αυτό που κάνει. Παρακαλώ, κύριε Νίλσον. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να διευκρινίσω πρώτα απ' όλα την έννοια. Το θέμα της ατομικής αξιολόγησης είναι το κατά πόσο η λεγόμενη ασφαλή χώρα είναι όντω ασφαλή για το συγκεκριμένο άτομο. Όχι το αν χρειάζεται διεθνή προστασία ή όχι ο ετών, μπορεί να τη χρειάζεται. Αλλά στην τρίτη αυτή χώρα που μπορεί να είναι η Τουρκία θεωρούμε κατά πόσο αν ο συγκεκριμένος είναι ασφαλής ή όχι. Αν διαπιστώσετε δηλαδή ότι το άτομο αυτό πράγματι χρειάζεται διεθνή προστασία και ότι μπορεί να έχει τέτοια πρόσβαση στην τρίτη χώρα, στην Τουρκία για παράδειγμα, τότε μπορείτε να πείτε ότι το αίτημα ασύλου είναι απαράδεκτο χωρίς να μπείτε στην ουσία και να επιστρέψετε το άτομο στην Τουρκία. Άρα υπάρχει πράγματι μια διάκριση ανάμεσα στο παραδεκτό ή όχι και στην εξέταση της ουσίας της αίτησης ασύλου. Όσον αφορά την Ελλάδα, εφαρμόζοντας την οδηγία, δεν έχουν πει ότι γενικά είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία, το κάνουν ατομικά κατά περίπτωση άρχισαν, αυτή τη βδομάδα ουσιαστικά να εφαρμόζουν την αρχή αυτή για όσους φτάνουν στα ελληνικά νησιά. Αυτό που απαιτεί οδηγία πάντως είναι ότι κάθε φορά η εξολόγηση γίνεται ατομικά, κατά πόσο δηλαδή για το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να έχει διεθνή προστασία στην τρίτη χώρα. Ακόμα δηλαδή και αν οριζόταν γενικά μια χώρα ως ασφαλής, πάλι θα έπρεπε να υπάρχει ατομικά η εκτίμηση για το συγκεκριμένο άτομο θεωρείται ασφαλής η χώρα ή όχι. Ο κύριος Δεπρέ. Συγγνώμη, ναι, θέλω... Εδώ νομίζω ότι βρισκόμαστε στο θέμα του εικονικού, γιατί υπάρχει μια πολιτική συμφωνία η οποία λέει ότι κάθε Σύριος υπήκος που θα ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα θα σταλεί πίσω στην Ελλάδα, λέει ο κύριος Δεπρέ και για κάθε έναν που πηγαίνει στην Ελλάδα θα επιστρέφεται ένας άλλος πίσω στην Τουρκία. Είναι συλλογικό αυτό, δεν είναι. Εσείς λέτε ότι ατομικά θα εξετάζονται, αλλά όλοι όσοι Σύριοι ζητούν άσυλο και το αίτημά τους θα θεωρηθεί παραδεκτό, θα επιστρέψουν στην Τουρκία. Δεν είναι συλλογική δράση αυτή. Δεν είναι ατομική. Ο κύριος Νιούτον είναι αλήθεια αυτό όσον αφορά τη συμφωνία. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία να γίνει ακριβώς αυτό. Αλλά για να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη, και αυτό το είπε και ο κύριος Γιούνκερ με δήλωσή του, ότι πρέπει να εφαρμόσετε το διεθνές δίκαιο, δηλαδή να τηρούνται τα κριτήρια τα οποία σας ανέφερα πριν, δηλαδή να επαληθεύονται κατά περίπτωση. Το δίκαιο υπερέχει. Και αυτό είναι αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών να κάνουν αυτή την αξιολόγηση και να εφαρμόζουν κατά περίπτωση το δίκαιο. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχουμε ολοκληρώσει την εμερήσια διαταξή για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστούμε για τη διερμηνία. Έχουμε δύο συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα. Μια έκτακτη την Δευτέρα 25 Απριλίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και μετά την 5η 28 Απριλίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιστροφή στα σπίτια σας.